Σας παρακαλώ να καθίσετε. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας. Iniziamo con eh, l'approvazione Ξεκινάμε με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Που φαντάζομαι ότι την έχετε στο φακελό σας. Εάν τώρα δεν υπάρχουν αντιρρήσεις ή άλλες παρατηρήσεις, και αυτή είναι η εντύπωση που έχω μπορούμε να θεωρήσουμε ότι εγκρίνεται αυτή η μέση διάταξη που φυσικά να τρέχει στην προηγούμενη προεδρία του κυρίου Ρόιλ, η διατύπωσή της. Δεύτερον, για τη σημερινή μέρα, έχουμε την, ε, τη διερμηνία σε όλες τις επίσημες γλώσσες του Κοινοβουλίου. Ε, το επόμενο θέμα είναι η έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της 10ης Νοεμβρίου 2011 που όπως ήθισε θα θεωρηθούν εγκεκριμένα τα πρακτικά αν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις ή σχόλια που θα διατυπωθούν μέχρι το τέλος της συνεδρίασής μας και εφόσον έχουμε την ψηφοφορία και δύο άλλα θέματα ε, συζήτησης στη συνέχεια, θα πρέπει να περάσουμε αμέσω στην παρουσίαση των κυρίων σημείων της μελέτης σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Έχουμε στη διάθεσή μας περίπου μία ώρα για την παρουσίαση αυτή και ξεκινάω τη συζήτηση για, ε, δίνοντας το λόγο στον δόκτορα Άλτμαν ο οποίος έχει 10 λεπτά για να παρουσιάσει τη μελέτη αυτή. Παρακαλώ, δόκτορα Άλτμαν. Mm, όχι, όχι, δεν θα μιλήσει, συγγνώμη, δόκτωρ Άλτμαν Όπως προβλεπόταν, αλλά προηγουμένως ο κύριος Μπρένικ Μέιερ θα λάβει το λόγο. Σας παρακαλώ λοιπόν να λάβετε το λόγο επί ένα δεκάλεπτο περίπου. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε για, το... για τη δυνατότητα που μου δίνετε να εκφραστώ ενώπιον των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λέγομαι Αντώνιος Μπρένικ Μέιερ και με τον κύριο Άλτμαν εκπροσωπούμε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που εξεπώνησε αυτή τη μελέτη η οποία σας έχει διαβιβαστεί και τις οποίες θέλουμε εδώ να παρουσιάσουμε τα κύρια σημεία. Πρόκειται για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανανεώσιμων Ενεργειών. Σε 10 λεπτά βέβαια είναι δύσκολο να παρουσιάσω μια μελέτη που εκτείνεται σε 150 σελίδες. 15 άτομα είναι η ομάδα η οποία συνέταξε αυτή τη μελέτη ή συνέβαλε στην εκπόνησή, της. Αυτό σας το λέω προκατακτικά. Σας φέρνω τώρα στο σκελετό της παρουσίασής μας. Θέλουμε να σας δώσουμε μια σύνοψη των περιεχομένων της μελέτης. Να δούμε μετά μερικά βασικά στοιχεία που είναι τα κύρια εμπόδια στην ανάπτυξη των δικτύων. για τη σχέση κόστους ε, ωφέλεια σε ό,τι αφορά τις επεκτάσεις των δικτύων, για τα θέματα προτεραιότητων στη διασύνδεση και περαιτέρω συστάσεις. Ξεκινώ λοιπόν με το περιεχόμενο της μελέτης. το βασικό πλαίσιο αυτής της μελέτης. Δεν νομίζω ότι θα δημιουργήσει εκπλήξεις σε εσά. Θέλουμε να έχουμε 20% ανανεώσιμες ενέργειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2020 και 80 95% μειώσεις σε εκπομπέ του άνθρωπος μέχρι το 2050, κάτι το οποίο απαιτεί και αλλαγές και μετασκευέ στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Η συμπερίληψη διακειμενόμενων πηγών ενέργειας δηλαδή ανανεώσιμων ενεργειών στο δίκτυο ηλεκτρισμού, ηλεκτρικής διανομής, στο... είναι κάτι το οποίο απαιτεί σημαντικές επενδύσεις. Ο στόχο τη μελέτη είναι να δούμε ποιε είναι οι αλλαγέ στι υποδομέ που χρειάζονται μέχρι το 2050, λαμβάνοντα υπόψη τι διάφορε προβλέψει για την ανάπτυξη των ανανεωσίμων ενεργειών. Δεύτερον, τα διάφορα σενάρια. Υπάρχουν διαφορετικά μάλλον σενάρια τα οποία βασίζονται σε διαφορετικέ παραδοχέ. Όλα αυτά όμως διατυπώθηκαν πριν από την καταστροφή της Φουκουσίμα και επομένως βασίζονται σε τέτοια δεδομένα πριν από την ε, καταστροφή αυτή. Δεύτερον, οι τεχνολογίες για την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων ενεργειών στο δίκτυο μπορεί να αλλάξουν φυσικά αυτή την εικόνα. Επίσης, αν δούμε τις προβλέψεις και τις προεκβολές δείχνουν οι αναλύσεις ότι μέχρι στιγμής τα πράγματα πηγαίνουν πιο γρήγορα από ό,τι προβλεπόταν. Είναι δηλαδή μεγαλύτερη επιτυχία στην ενσωμάτωση των ανανεωσίμων ενεργειών. Κάτι ακόμα το οποίο είδαμε είναι οι ήδη δημοσιευμένες προτεραιότητες για ανάπτυξη υποδομών η σχέση κόστους και ωφέλεια σε σχέση με τις υποδομές, θα επαναληφθούμε στο θέμα αυτό, που υπογραμμίσω τη σημασία του. Θέλω να τονίσω και τη δυσκολία του να έχουμε σαφή αξιολόγηση αυτή αυτής της σχέσης, τους στόχους πολιτικής και την νομοθεσία των κρατών μελών και τα προσκόμματα για την σύνδεση των ανανεώσιμων ενεργειών με το δίκτυο. Πιστεύω ότι οι συστάσεις μας και τα πορίσματά μας είναι πράγματι ε, πλήρη και εκτενή. Έρχομαι στην επόμενη διαφάνεια και εδώ αναφέρω μερικές από τις κύριες μέρημνες μας. Τις ονομάζουμε κύριες μέρημνες γιατί θεωρούμε ότι θα πρέπει αυτό να σας μείνει μετά από την παρακολούθηση αυτής της παρουσίασης. Πρέπει να μείνει στη μνήμη σας. Όπως σας είπαμε, η σε αυτή ανάλυση σχέσης κόστους ωφέλειες σε σχέση με τα σχέδια υποδομών <clears throat> τα δυνητικά ωφέλη και οι δυνητικές συγκρούσεις που μπορούν να προκύψουν για την εσωματώση στην αγορά ενέργειας και την ασφάλεια της τροφοδοσίας με ηλεκτρισμό. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε περαιτέρω ότι η βελτίωση, η ανάπτυξη των υποδομών δικτύου και των διασυνδέσεων θα οδηγήσει, ε, θα οδηγήσει σε καλύτερη <clears throat> κυκλοφορία <clears throat> των προϊόντων ενέργειας, θα έχουμε λιγότερη εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα, ενδεχομένω θα έχουμε βιοκαύσιμα, μπορεί να έχουμε, ε, να έχουμε εισαγωγές ηλιακής ενέργειας και τίθεται και το θέμα των σπανίων γεών που έχει να κάνει με τη χρήση των, με την αξιοποίηση των ανανεώσιμων ενεργειών. Θα υπάρξουν επομένως και επιπτώσεις <clears throat> στην τιμολόγηση της ενέργειας που θα είναι και διαφοροποιημένες ενδεχομένως οι τιμές της ενέργειας ανάλογα με την περιοχή. Ε, μια μεγάλη πρόκληση θα είναι όχι μονάχα η εξισορρόπηση του, του, της παροχής από το δίκτυο για την αντιμετώπιση της ζήτησης, αλλά και η ανάγκη να υπάρχει και αποθεματική παροχή ηλεκτρισμού για να αντιμετωπίσει εχμές ηλεκτρισμού και αυτό φυσικά αυξάνει το κόστος της δημιουργίας υποδομών. Αν δούμε τώρα και τα αποτελέσματα που θα προκύψουν για το περιβάλλον των νέων αυτών υποδομών, μπορούμε να βούμε σε περισσότερη λεπτομέρεια για τα θέματα αυτά, αλλά σε ό,τι αφορά τις πολιτικές οι οποίες θα πρέπει να ακολουθηθούν, θα πρέπει να δούμε πώς συνδέεται η πολιτική αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των μηχανισμών εμπορίας εκπομπών ως πηγές υποστήριξης της ανάπτυξης ανανεώσιμων ενεργειών, γιατί μπορεί να υπάρχουν στοιχεία τα οποία οδηγούν σε συγκρούσεις και τριβές. Θα εξετάσουμε επίσης στη μελέτη αυτή τα διάφορα προσκόμματα, πιο λεπτομεριακά σε ό,τι αφορά την κοινωνική, οικονομική ή διοικητική τους φύση. Και θα δούμε και ποιος είναι ο λόγος των λιπτών αποφάσεων ώστε να εξασφαλίσουμε ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε την, ε, τους στόχους μας επικαιροποιώντα την πολιτική για την ανανεώσιμη ενέργεια και τις υποδομές της. Κάτι το οποίο είναι σαφέ είναι ότι έχουν γίνει ήδη πολλά πράγματα για να προετοιμαστούμε για αυτέ τι αλλαγέ. Υπήρξε σημαντικό συντονισμό στα θέματα αυτά. Αυτό όμω το οποίο θα είναι απαραίτητο περαιτέρω είναι όχι μόνο ο συντονισμό αυτό καθεαυτό, αλλά και η ανάληψη ευθυνών από του λήπτε αποφάσεων. Ίσως έχετε ξαναδεί τις επόμενες, τα, τις επόμενες εικόνες που δείχνουν ποια είναι η γεωγραφική κατανομή των πηγών αιωλικής και ηλιακής ενέργειας. Αριστερά είναι η αιωλική πόρη, δεξιά είναι η ε, ακτινοβολία, η ηλιακή ακτινοβολία η οποία προσπίπτει σε κάθε περιοχή της Ευρώπης. Βέβαια δεν είναι προβλέψιμες οι πηγές αυτές, δεν είναι προβλέψιμη η ύπαρξη ανέμου, η, η Και αυτό θα πρέπει να μας οδηγήσει σε κάποιες ε, αλλαγές στο σύστημά μας για να ενσωματώσουμε και αυτές τις πηγές ενέργειας. Αυτό το οποίο θετικό είναι ότι αυτές οι πηγές μπορούν να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες μας. Αλλά δεν μπορεί να επιτευχθεί αυτό με τις τωρινές υποδομές. Οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν προκύπτουν από το γεγονό ότι είναι διακειμενόμενες πηγές ενέργειας αυτέ οι ανανεώσιμε ενέργειες, δεν είναι πάντα διαθέσιμες, δεν είναι διαθέσιμες όταν τις χρειαζόμαστε. Υπάρχει ανάγκη λοιπόν μεταφοράς ενέργεια των ανανεώσιμων ενεργειών από τον τόπο παραγωγής του στον τόπο κατανάλωσης και αυτό αφορά και τη χαμηλή τάση και την υψηλή τάση αλλά και τη μεσαία τάση. Υπάρχει Βλέπετε στο διάγραμμα αυτό τις άλλες δύο πηγές ανανεώσιμης ενέργειας, την ε, γεωθερμία και το υδροηλεκτρικό δυναμικό που επίσης είναι άνισα κατανεμημένα στην Ευρώπη. Πιο, πιο ελαφρύ χρώμα στα υδροηλεκτρικά σημαίνει μεγαλύτερο δυναμικό. Όπω είπα, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ισορροπήσουμε τη ζήτηση με την προσφορά, πρέπει να σταθροποιήσουμε τα επίπεδα ζήτηση και από την άλλη να υπάρχει ευελιξία στην παραγωγή. Οι διακυμάνσεις δεν είναι μόνο σε καθημερινή αλλά και σε εποχιακή βάση. Οπότε, τι αλλαγές αναμένουμε να γίνουν. Προφανώς η επέκταση του δικτύου μετάδοσης είναι μια δυνατή επιλογή για να διευκολύνουμε την ε, διασύνδεση της ανανεώσιμης ενέργειας, επιτρέποντας την συνεχή εξορρόπηση της ε, προσφοράς με τη ζήτηση, αλλά πρέπει να συμπεριληφθούν και άλλες επιλογές, όπως η αλλαγή του σχεδιασμού της αγοράς, η ε, διαχείριση της προσφοράς, η μετατροπή του ηλεκτρισμού σε τελική ενέργεια για άλλες χρήσεις και εδώ πέρα μιλάμε για μεταφορές, θέρμανση και βιομηχανικές χρήσεις, αντίδραση στην ε, ζήτηση και αποθήκευση ενέργειας. Και αποθήκευση ενέργειας νομίζω θα μας απασχολήσει ε, νομίζω αργότερα. Υπάρχουν και απαιτήσει για απέτηση για ε, αποθήκευση αποθεμάτων πετρελαίου και αερίου. Πρέπει να σκεφτούμε και τα αποθέματα ηλεκτρισμού. Η επόμενη διαφάνεια σας δίνει μια ιδέα των διαφόρων επιλογών. Ο κάθετος άξονας ε, ε, οριζόντιος, με είναι η αύξηση του ποσοστού των διαφόρων πηγών παραγωγής ε, και ο κάθετος άξονας είναι το κόστος. Προσπαθούμε δηλαδή να δούμε το ποιο θα είναι το κόστος, αν θα έρθουν όλα μαζί, αν έχουμε μια σταδιακή εισαγωγή τους και σε ποιο κόστος ελπίζουμε και αναμένουμε να γίνουν αυτά τα πράγματα. Πρέπει να πούμε κάποια πράγματα. Όλες αυτές οι επιλογές ήδη συμβαίνουν με τη μία μορφή ή την άλλη ε, σε ένα βαθμό. Και το ιδεώδες μείγμα λύσεων θα εξαρτηθεί από τις τοπικές συνθήκες. Καμιά φορά είναι κανείς κοντά σε μία λύση αποθήκευσης, άλλες φορές όχι. Μία πανευρωπαϊκή προσέγγιση χρειάζεται για να έχουμε μία πανευρωπαϊκή πολιτική με τρόπο αποτελεσματικό. Γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη την οικονομική βιωσιμότητα των εμπλεκομένων εταιριών και όσων έχουν βεβαίω συμφέρον. Βλέπουμε λοιπόν να σας πούμε τι μπορείτε να βρείτε στην μελέτη, ας πούμε, στις λεπτομέρειες. Έχουμε εδώ πέρα τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες εμποδίων. Αυτό το οποίο έχουμε δει εδώ πέρα είναι πως ε, τα τεχνικά εμπόδια, τα έχουμε τελευταία βεβαίως, ε, είναι τα πιο εύκολα και αυτά που είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμα. Ε, τα άλλα τρία τα διοικητικά, κοινωνικά και οικονομικά προσκόμματα είναι αυτά τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν και θα χρειαστεί πολιτική βούληση σε επίπεδο ένωσης και κρατών μελών. Αποφασίσαμε ε, πως η κατάταξη δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία καθώς το καθένα από αυτά μπορεί να έχει σημασία διαφορετική ανάλογα με τα τοπικά χαρακτηριστικά του κάθε Επειδή ο χρόνος πιέζει, θα δώσω τον λόγο στο Ματίας σε λίγο. Και για να σας δείξω εδώ πέρα τις διαφάνειες όσον αφορά την στρέβλωση της αγοράς, τα διασυνοριακά ζητήματα αν έχουμε δύο ή περισσότερες χώρες, ε, τα αντικίνητρα επένδυσης ε, για τους διαχειριστές του δικτύου διανομής που δεν μπορούν να ανακτήσουν το κόστος και την έλλειψη ιδιωτικής ε, χρηματοδότησης καθώς και τις διοικητικές διαδικασίες και τις αβεβαιότητες για το μέλλον. Τα κοινωνικά εμπόδια είναι οι περιβαλλοντικές ανησυχίες, καθώς ε, ε, υπάρχουν προβλήματα π.χ. για τις γραμμές υψηλής τάσης. Τα ζητήματα υγείας δεν έχουν μέχρι στιγμής εξεταστεί και πρέπει να τα δούμε πολύ προσεκτικά όσον αφορά την επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους και βεβαίω ο αρνητικός αντίκτυπος στο τοπίο ε, που μπορεί βεβαίως να μειώσει και τις αξίες της γης. Όσον αφορά τα διοικητικά εμπόδια, έχουμε εθνικού κανονισμούς που μερικές φορές είναι αντίστοιχοι με του ευρωπαϊκούς, διαδικασίε αδειοδότηση μακροσκελή. Ε, η πρόσβαση στο δίκτυο είναι αργότερη από την παραγωγή ε, από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και υπάρχει και η μελέτες περιβαλλοντικού αντικτύπου που είναι αυτή τη στιγμή πολύ μακροσκελής και περιορίζουν ε, και επίσης κοστίζουν πάρα πολύ. Θα δώσω τώρα τον λόγο στο Ματίας για να καλύψει τα υπόλοιπα στοιχεία της ε, παρουσίασής μας. Ευχαριστώ. Θα εστιαστώ τώρα αφενός σε μία ανάλυση κόστους οφέλους για τις υποδομές ηλεκτρισμού και στις προτεραιότητες που συζητάμε αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις υποδομές αυτές. Ποιος είναι ο στόχος ε, των αναλύσεων κόστους κόστους-οφέλους για να μας υπενθυμίσει γιατί είναι σημαντικό αυτό το ζήτημα. Στόχο έχει να κατευθύνει την επιλογή επενδύσεων και την κατανομή του κόστους στους ενδιαφερομένους. Αυτό σημαίνει όχι μόνο έγκριση ή μη έγκριση προτινόμενων έργων, αλλά επίσης να βρούμε ποια από αυτά παρουσιάζουν το μεγαλύτερο όφελος ε, σε σχέση με το κόστος. Ένας τρόπος δηλαδή κατάταξης βαθμολογίας των έργων. Και να σας υπενθυμίσω επίσης το ότι η ανάλυση κόστους οφέλους καλύπτει όλες τις πτυχές ε, της υποδομής, όχι μόνο τις ανανεώσιμες. Θα το έχετε δει αυτό το διάγραμμα φαντάζομαι στο παρελθόν. Δίκτυο, ε, οι επενδύσεις στο δίκτυο γίνονται για τρεις λόγους. Για να έχουμε ασφάλεια παροχής ε, ενέργειας, για να ενσωματωθούν οι ανανεώσιμες πηγές και για να ε, ενσωματωθούν και να ολοκληρωθούν οι ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρισμού. Το τι κοιτάμε τώρα είναι τέσσερις ε, διαφορετικοί τύποι υποδομών. Ένα, το σημαντικότερο βεβαίω είναι η επέκταση του δικτύου, αλλά μιλάμε επίσης για αποθήκευση, κάτι το οποίο συμπληρώνει βεβαίως την επέκταση αυτή και κάποιες επεκτάσεις μπορεί να μην ε, χρειάζονται στην περίπτωση που μπορούμε να αυξήσουμε την αποθηκευτική δυνατότητα. Επίση, η αντίδραση στη ζήτηση μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην ενσωμάτωση των ανανεώσιμων και μπορεί να μειώσει την ανάγκη για περαιτέρω δίκτυα. Η διαχείριση της συζήτηση είναι επίσης ένα θέμα που θα μπορούσε να παίξει ένα πιο σημαντικό ρόλο από ό,τι παίζει σήμερα. Ένα σημαντικό ζήτημα που πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι πως ε, για να αποσβέσουμε το κόστος της υποδομής ε, χρειάζονται δεκαετίες. Μπορεί να πάμε πέρα από το 2050 για ό,τι αποφασίσουμε σήμερα. Και βεβαίως το άλλο στοιχείο είναι πως χρειάζεται ίσως μια δεκαετία ή και παραπάνω για να ε, εφαρμοστούν ε, τα έργα αυτά. Μιλάμε λοιπόν για μεγάλο χρόνο κατασκευής και ζωής για να γίνει μια σωστή ανάλυση κόστους κόστους-οφέλους. Υπάρχουν λοιπόν πολλές αβεβαιότητες που σχετίζονται με μια ανάλυση κόστους κόστους-οφέλους. Κόστος και όφελος είναι δύσκολο να υπολογιστεί με βεβαιότητα, ειδικά όταν μιλάμε για μακροπρόθεσμα ζητήματα. Ποιος ξέρει ποιο θα είναι το κόστος και το όφελος το 2050. Είναι δύσκολο αυτό. Έχουμε κάποιες άλλες παραμέτρους ε, από τις οποίες εξαρτώνται τα αποτελέσματα, δηλαδή τιμές των καυσίμων, προφανώς, το κόστος των επενδύσεων αυτών, η αξία της ασφάλειας του συστήματος, ε, συνθήκες λειτουργίας κτλ. Τι κάνουμε λοιπόν με αυτές τις αβεβαιότητες. Το σημαντικό είναι να έχουμε διαφορετικά σενάρια. Όχι μόνο δύο ή τρία, αλλά πολλά σενάρια. Ας πούμε 10, 15, 20 και μετά να δούμε τι μπορεί να είναι μια σωστή απόφαση επενδύσεων που θα προκύψει από διάφορα σενάρια και σημαντικό είναι να υπάρχει και μια ανάλυση ευαισθησίας ανάλογα με τις διακυμάνσεις των διαφόρων σενάριων και το τι θα επηρεάσει περισσότερο το κόστος και το όφελος. Τα βασικά ωφέλη είναι αρκετά μεγάλος ο κατάλογος τώρα, δεν θα τα αναφέρω όλα. Είναι πως επί της αρχής υπάρχει άξιση στην αποτελεσματικότητα της χρήσης των ανανεώσιμων, μείωση του κόστους λειτουργίας του συστήματος, αύξηση του επίπεδου ανταγωνισμού, αυτό σχετίζεται κυρίως με την ε, ολοκλήρωση της αγοράς ηλεκτρισμού, αύξηση στο επίπεδο της ασφάλειας ε, προμήθειας ενέργειας, καθώς μπορούμε να δώσουμε την ενέργεια από ανανεώσιμε και σε χώρε εκτό συνόρων κτλ. Επίση, αυξάνεται η ευρωστία τη αγορά και διαχείριση επίσης της ζήτησης. Η αύξηση της αποτελεσματικότητας ε, της αποθήκευσης ενέργειας επίσης ενισχύεται και πρέπει να πω εδώ πέρα πως το επίπεδο αποθήκευσης του ηλεκτρισμού στην Ευρώπη είναι εξαιρετικά χαμηλό σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη πηγή ενέργειας. Π.χ. η αποθήκευση φυσικού αερίου είναι διαφορετική τάξη μεγέθους. Οπότε η αποθήκευση του ηλεκτρισμού είναι πολύ πιο δύσκολη από οποιαδήποτε άλλη μορφή ενέργειας, γι' αυτό έχουμε πολύ χαμηλό επίπεδο αποθηκευτικής δυνατότητας στην Ευρώπη και τέλος υπάρχει πιθανή αύξηση στο μήθος και την αποτελεσματικότητα των νέων παραγωγών λόγω της αύξησης του μεγέθους της αγοράς. Ποια είναι τα αποτελέσματα τώρα της ε, ανάλυσής μας όσον αφορά τις υφιστάμενες δομές. Η ανάλυση δείχνει πως θα έχουμε υψηλότερο όφελος από κόστος, αλλά πρέπει να υπολογίσουμε ακριβώς το κόστος και το όφελος, όπως είπα, εφαρμόζοντας διάφορα σενάρια να δούμε το τι είναι πιο εύρωστο και τι όχι. Οπότε τα ωφέλη είναι πολύ περισσότερα από την αύξηση των ανανεώσιμων αλλά δεν θα διανεμηθούν εξίσου σε όλους. Οπότε η ανάλυση κόστος ωφέλους θα μπορέσει να κατανείμει το κόστος στους διάφορους ενδιαφερομένους. Τώρα, αν δείτε την ανάλυση κόστος ωφέλους για τις προτεραιότητες ε, στις επενδύσεις. Αυτές είναι οι προκλήσεις που έχουμε. Οι στόχοι του εθνικού σχεδίου ε, δράση. Με κάποιες χώρες, Ιρλανδία, Δενία, Ελλάδα, Ισπανία κτλ. θα έχουν μεγάλα ποσοστά κειμενόμενων ανανεώσιμων στο δίκτυο και Έχουμε το εθνικό επίπεδο και από την άλλη έχουμε και τις απόλυτες τιμές ε, παραδείγματο χάρη αιωλική ενέργειας στο γαλλικό δίκτυο. Το μεγαλύτερο απόλυτο λοιπόν είναι σε Ισπανία, Πορτογαλία, ε, ε, Γερμανία και Ελλάδα ας πούμε. Αυτές είναι οι προκλήσεις. Τι σημαίνει αυτό για το δίκτυο. Έχουμε προτείνει προτεραιότητες στο ενεργειακό πακέτο υποδομής που προκρίθηκε τον Οκτώβριο, προτάθηκε με τον Οκτώβριο, καθώς επίσης και το ΕΝΤΣΟΗ e. Αυτά προτάθηκαν. Η βασική κριτική λοιπόν βασί, είναι στο ότι βασιζόμαστε σε μια λογική από κάτω προς τα πάνω, δηλαδή κάθε χώρα υποβάλλει αυτό το οποίο θεωρεί ότι είναι το σημαντικότερο έργο, αλλά δεν υπάρχει μια προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω, από ευρωπαϊκή προοπτική, δηλαδή αν δούμε την Ευρώπη από το διάστημα χωρίς σύνορα, ποια θα πρέπει να είναι η ε, προτεραιότητα. Δεν υπάρχει λοιπόν τέτοια λογική, αλλά πηγαίνουμε προς τα εκεί. Εάν δείτε λοιπόν το άρθρο 12 του πακέτου υποδομών, της πρόταση των Ευρωπαϊκών Δικτύων Ενέργειας ε, λέει πως ε, η ΕΝΣΟΗ πρέπει να προετοιμάσει μια μεθοδολογία για μια ενιαία ανάλυση κόστους κόστους-οφέλους για την ενέργεια σε ολόκληρο το σύστημα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για έργα κοινού συμφέροντος. Θεωρούμε πως είναι φιλόδοξο να αναμένουμε η ΕΝΣΟΗ να υποβάλει αυτή τη μεθοδολογία μόλις ένα μήνα μετά τη θέση ενισχύ του προτινόμενου κανονισμού. Υποθέτουμε πως για να υπάρχει μια σωστή μεθοδολογία θα απαιτηθεί περισσότερος χρόνος. Παρά το ότι έχει γίνει κάποια ανάλυση κόστους ωφέλους θεωρούμε πως αυτές οι οποίες έχουν γίνει μέχρι στιγμής δεν καταλήγουν κάπου όσον αφορά το εάν είναι βέλτιστες οι, προ... οι προτεραιότητες που έχουμε αυτή τη στιγμή και δεν έχουν φτάσει ακόμα στο βαθμό λεπτομέρειας και ευρωστίας που θα θεωρούσαμε ικανοποιητικό από επιστημονική και πολιτική σκοπιά. Αν δούμε το δίκτυο Βλέπετε το επίπεδο διασύνδεσης που υπάρχει. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια και βλέπουμε πού είναι οι προτεραιότητες σύμφωνα με το πιλωτικό δεκαετές σχέδιο. Αυτή θα είναι η κατάσταση δηλαδή 2020 με βάση τον σχεδιασμό και βλέπουμε πως παρά το ότι Μοιάζουν ε, πάρα πολύ καλές αυτές οι προτάσεις, δεν υπάρχει επιστημονική βάση για να πούμε αν είναι ή όχι. Οι ερευνητικέ λοιπόν απαιτήσει σημαίνει πως θα πρέπει να μπούμε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό λεπτομέρειας και να υπάρχει μια συνεκτικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό μας λέει λοιπόν αυτή η διαφάνεια. Τώρα ας περάσουμε στην τελευταία διαφάνεια οι συστάσεις. Σημαίνει πως οι υποδομές θα πρέπει να έχουν ένα μεγάλο βαθμό υποκατάστασης, δυνατότητας υποκατάστασης, δηλαδή ο αριθμός εναλλακτικών για κάθε έργο το οποίο προτείνεται και ανάλυση κόστους ωφέλους θα πρέπει να γίνει για κάθε ένα από αυτά για να δούμε ποια είναι τα βέλτιστα από πλευράς κόστους. Πολλαπλά σενάρια, όπως είπαμε, χρειάζεται να εξεταστούν γι' αυτό και να δούμε τα πράγματα μακροπρόθεσμα γιατί οι υποδομές αυτές θα λειτουργούν οι περισσότερες μέχρι το 2050. Όπως είπα, το επίπεδο έρευνας πρέπει να αυξηθεί για να υπάρχει ευρωστία στις μεθόδους και τα αποτελέσματα ως βάση για τις πολιτικές αποφάσεις. Νομίζω πρέπει να σταματήσω κάπου εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και είμαστε στη διάθεσή σας να απαντήσουμε ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε θερμά και τους δύο και δίνω το λόγο στον κύριο Κορεάτη Κάμπος για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. και ευχαριστώ θερμά για, τον, για το γενναιόδωρο χρόνο που μου δώσατε. Ξεκινώ ευχαριστώντας και συγχαίροντας τους ε, συντάκτες της εκθέσεως που κρίνω πολύ σημαντική γιατί μπορεί πράγματι να βοηθήσει στην εκτέλεση του κανονισμού χάρη στην πρακτική έρευνα και την ανάλυση του κόστους ε, και της αποτελεσματικότητας. Έχω μια σειρά από Πρώτον, σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως οι δυσκολίες ή καλύτερα τα εμπόδια που υφίστανται αυτή τη στιγμή ή στο περιβάλλον ή φυσικά εμπόδια για την ανάπτυξη ε, δικτύων onshore. Σε ποιο βαθμό λοιπόν πιστεύετε ότι τα εμπόδια αυτά περιβαλλοντικού, οικονομικού, τεχνικού, κοινωνικού χαρακτήρα που καθιστούν ε, ε, διπλάσιο το κόστος ε, του onshore δικτύου σε σχέση με το offshore, θεωρείται ότι πράγματι αιτιολογούν αυτό, αυτή την τιμή. Μην με ρωτήσετε που βρήκα το, τη διαφορά αυτή στην, στο κόστος. Ε, εν πάση περιπτώσει διπλάσιο κόστος βλέπω από τις πηγές μου, μάλιστα υπάρχουν πηγές που αναφέρουν και τετραπλάσιο κόστος. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε λοιπόν ότι ενδέχεται να παρεμποδίσουν την ρευστότητα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σε ποιο βαθμό οι επικρίση αυτές ως προς την επιλογή του προτύπου που θα επιλεγεί, τεχνολογία αποθήκευσης, και το, η μεγάλη απόσταση που έχουμε βεβαίως διανύσει σε σχέση με τις τεχνικές πρόοδους, ε, παρόλα αυτά καθιστούν, αφήνουν ως μόνη τη δυνατότητα την αποθήκευση ε, ε χώρες οι οποίες δεν διαθέτουν τεχνολογία αποθήκευσης και πρέπει να μεταβούν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ε, αντιμετωπίζουν πολύ περισσότερες δυσκολίες από εκείνες τις χώρες οι οποίες έχουν το λεγόμενο καλό υδρικό μείγμα. Πιστεύετε λοιπόν ότι θα μπορέσουμε στα προσεχή χρόνια να εξασφαλίσουμε επαρκείς ε, τεχνολογικές δυνατότητες ώστε να αποθηκεύσουμε την ε, ε, ενέργεια που υφίσταται φερρυπίν από υδρογόνο και από τα φωτοβολταϊκά. Γιατί δεν ακούω να μιλάτε για, τα, για την ενέργεια χάρη στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Ε, ξέρω ότι έχει ίσονα ε, αναλογία. Αλλά παρόλα αυτά θα παραμείνει πτωχός συγγενής του συστήματος ή του νέου καθεστώτος. Γιατί γνωρίζω βεβαίως ότι έχουν λιγότερη επίπτωση στο περιβάλλον τέτοιου είδους τεχνολογίες, φερρυπίν, στις οικιακές χρήσεις. Και τέταρτη ερώτηση. Διατυπώθηκε ανεπικρίσεις σε αυτές τις προτάσεις ε, αρκετές φορές στην πατρίδα μου γιατί ε, πάντα φαίνονται όλα αυτά πολύ ωραία αλλά εν τέλει την επένδυση στις νέες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ε, καλύτερα την πληρώσει ο καταναλωτής. Και ξέρουμε μερικές φορές ότι αυτές οι επενδύσεις πολλές φορές είναι ιδιαίτερα ε, δαπανηρές. Και όπως και να προβάλλεται τελικά η κατάσταση, ξέρουμε ότι τελικώς ε, στο τέλος αυτής της ιστορίας, αυτός που θα κληθεί να βάλει το χέρι στην τσέπη, είναι ο καταναλωτής. Ό,τι και να λέμε. Υπάρχει λοιπόν εναλλακτική. Επίσης, ως προς το κόστος και το αποτέλεσμα, ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολο βέβαια να προσμετρηθεί ε, σε όρους επακριβής το ε, οτιδήποτε έχει να, κάνει, να, να έχει να κάνει με ακίνητα. Αλλά πιστεύετε ότι θα μπορούσε η ΕΝΣΟ και η ΕΣΕΡ να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρουν τέτοια σχέδια και για το μέλλον. Πιστεύετε ότι ενδεχομένως χρειαστεί να αλλάξει η μέθοδος υπολογισμού ε, του κόστους. Εν πάση περιπτώσει, σε ποιο βαθμό μπορεί να συμβάλλει όλο αυτό. Και σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι μπορεί να αξιοποιηθεί η τεχνολογία αυτή ή θεωρείτε ότι είτε οι διαχειριστές είτε αυτοί που θα κληθούν να εκτελέσουν αυτές τις ε, ε μεθόδους στο μέλλον θα μπορέσουν να το πράξουν ικανοποιητικά. Ευχαριστώ πολύ. Η Πρόεδρος, δύο λεπτά για τους λοιπούς συναδέλφους που έχουν ζητήσει το λόγο. Κύριος Αντώ είναι ο πρώτος. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πολύ τους, τους κύριους που Αναφέρατε ένα πολύ σημαντικό σημείο, ότι δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, διαπραγματευόμαστε και προσδιορίζουμε ένα νέο κανονισμό που πιστεύουμε θα ε, προσφέρει νέα κριτήρια και αναλύσεις, όπως εσείς άλλωστε αναφέρατε για το πώς αναλύσεις και το καθεξής που επίσης όμως θα πρέπει να ε, παραγάγει εν τέλει και κοινά ε, εγχειρήματα, ε, σχέδια για κοινά έργα. Αυτή τη στιγμή όμως φαίνεται ότι τα όποια σχέδια υπάρχουν είναι μόνο εθνικού χαρακτήρα. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να σχεδιάσουμε μια διαδικασία η οποία άπαξ και προσδιοριστούν τα κριτήρια, οι δείκτες γίνουν οι αναλύσεις, θα μας επιτρέψει να στραφούμε προς τα κράτη και να πούμε, κοιτάξτε, 27 χωριστά εθνικά σχέδια δεν είναι απαραίτητα προς όφελος, προς το κοινό όφελος, ούτε και είναι αποτελεσματικότερα. Γι' αυτό λοιπόν και ίσως η επολογία αυτή τη στιγμή να είναι εσφαλμένη, γιατί ίσως να προσδιορίζονται περισσότερο σχέδια εθνικού ή διεθνικού χαρακτήρα, διμερούς καλύτερα χαρακτήρα, ενώ η Ευρωπαϊκή Ενωσιακή ευρωπαικη ενωσιακη διεσταση ε, χάνεται. Και ενώ η επένδυση που θα γίνει για τις ε, υποδομές αυτές πιστεύω θα μπορούσε να δώσει πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Καλώς λέει η Πρόεδρος, κλείνω τον κατάλογο των ε, μιλητών. Διαφορετικά θα προλάβουν οι συνάδελφοι να απαντήσουν. Ο κύριος ε, Αλμπερτίνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε και αν μου επιτρέπετε να κάνω μια ερώτηση λίγο εκτός θέματος Ζητώ συγγνώμη λοιπόν προκαταβολικά, αλλά με την ε, μελέτη αυτή την οποία είδαμε μόλις σήμερα και εδώ και καθώς είμαι και νέος στην Επιτροπή, ίσως κάνω κάποιο ατόπιμα. Στο συγγνώμη προκαταβολικά. Θα ήθελα να πω λοιπόν ότι ασχολούμαστε ως το δυνατόν πιο αντικειμενικά για την παραγωγή, την διανομή της ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές και εσείς βέβαια ε, αναφερθήκατε στις πιο κλασικές, αιωλική, γεωθερμική, ηλιακή κτλ. Εγώ διατέλεσα για πολλά χρόνια δήμαρχος του Μιλάνου και από τις ε, πιο χρήσιμες ανανεώσιμες πηγές θα έλεγα ότι θεωρώ εκείνες που απορρέουν από τους τόνους των αποβλήτων που συσσωρεύονται στις χωματερές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάνω από το 80% του πληθυσμού των χωρών μας ζει σε αστικά κέντρα και έτσι θεωρώ ότι έχουμε με το δεδομένο αυτό μια πολύ σημαντική πηγή ενέργειας. Με την αποτέφρωση ε, και τους ε, ε, τις μονάδες αυτές καύσης που μπορούν να παράσχουν πολύ μεγάλη ε, υπηρεσία και για το περιβάλλον και για την ενέργεια και για την οικονομία ασφαλώς γιατί κοστίζει πολύ ακριβά η ε, καύση, η αποτέφρωση των σκυβάλων ε, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να κερδίσουμε πολλά. Δεν το αναφέρατε όμως αυτό και επιτρέψτε μου να υποβάλω στην κρίση σας και αυτή την ε, διάσταση που ενδεχομένω να αξίζει και χωριστή έκθεση. Επίσης, μια άλλη παρατήρηση, κάποιοι επιστήμονες, που ίσως δεν είναι θεόπνευστοι, θεωρούν ακόμη ότι οι πυρηνικές μονάδες με τεχνολογία που αναμένεται να αναπτυχθεί σε καμιά δεκαετία χρόνια, δεν θα χρησιμοποιούν πλέον ως καύσιμο ουράνιο από ορυχεία, αλλά ουράνιο από την θάλασσα αντλούμενο, ε, δεδομένου ότι το ουράνιο είναι παρόν ε, παντού στο, στην Ιφίλιο, νομίζω ότι θα είναι εύκολο αυτό και έτσι μπορούμε να μιλούμε πλέον και για ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Ο κύριος Πρόντι. Ευχαριστώ πρόεδρο. Μόλις τώρα είδα την έκθεση και στο συγγνώμη για οποιοδήποτε ατόπιμα, αλλά βλέπω ότι απουσιάζει μία συζήτηση πολύ σημαντική που αφορά τα super grid, δηλαδή τις ε, δομές αυτές ε, διαρκούς υψηλής τάσης, οι οποίες ασφαλώς χρειάζονται χρειάζεται να ληφθούν υπόψη γιατί έχουν ε, χαμηλότερες απώλειες, κατά τρεις φορές χαμηλότερες απώλειες από τα λοιπά δίκτυα. Νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό μπορούμε να αξιοποιήσουμε πολύ καλύτερα τις ανανεώσιμες, ε, να αντισταθμίσουμε μάλλον τις ε, ε χάρη ανανεώσιμες ε, πηγές και όταν λέω αντιστάθμιση εννοώ ε, μια μελέτη συγκριτική των διαφόρων πηγών ενέργειας ε, που θα οδηγούσε σε λύσεις πολύ πιο ενδιαφέρουσες από την αποθήκευση γιατί θα μας επέτρεπε ήδη ε, η φυστάμενη ενέργεια να την αξιοποιούμε πολύ πιο σωστά. και έτσι η πιο πολύτιμη εκδοχή της ενέργειας, η πιο πολύτιμη μορφή της ενέργειας, δηλαδή η ηλεκτρική ενέργεια θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στο βέλτιστο. Και μια και ο συνάδελφος μίλησε για απορρίμματα, θα πρότεινα και εγώ την διάσταση της βιομάζας. Γιατί να μην αποθηκεύουμε τη βιομάζα αντί να προσπαθούμε να αποθηκεύουμε ηλεκτρική ενέργεια. Το υδρογόνο μπορεί να αποθηκευτεί πριν να μετατραπεί σε ηλεκτρική ενέργεια, αφού υπάρχει δυσκολία με την ηλεκτρική ενέργεια. Ευχαριστώ κύριο Σκέλη. Ευχαριστώ πολύ. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους δύο μελίτες, ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι παρουσιάσεις τους. Ε, δύο παρατηρήσεις, το 2020 ασφαλώς ε, σαν στόχος παραμένει ενισχύει, είναι πάρα πολύ σημαντικός και μάλλον μέχρι να ξεκινήσουν ε, τα μεγάλα αυτά σχέδια να έχει πια εκπνεύσει και η δεκαετία που μας χωρίζει πλέον από το στόχο αυτό. Όμως ήθελα να βερθώ και στην αποθήκευση ενέργειας και τη γενικότερη στρατηγική που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε. Επίσης, σε ποιο βαθμό είναι απαραίτητη μια προσέγγιση από άνω προς τα κάτω. Και διοικητικά εμπόδια που ενδεχομένως υπάρχουν, πώς θα μπορούσαν να ε, εξαλειφθούν. Ίσως θα ήταν καλό να κοιτάξουμε την ευρωπαϊκή ε, διάσταση ως βάση για τα δίκτυα αυτά. Και η οικονομική κατάσταση ξέρουμε ότι μας υποχρεώνει να προχωρήσουμε και για λόγους ε, δημοσιονομικούς σε συνεργασία. Επίσης, εάν ε, αληθεύουν κάποιες αναφορές που αφορούν ε, τις πρόοδους της Ρωσίας ως προς την τεχνολογία ε, στον τομέα αυτών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο κύριος Τούρμες. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω πώς φτάνουμε στο συντονισμένο αυτό σχεδιασμό των δικτύων και από άνω προς τα κάτω και από κάτω προς τα άνω. Και για να συμπληρώσω τόσο ακούστηκαν νωρίτερα, θα έλεγα ότι είναι πολύ δύσκολο να εξασφαλίσουμε πρόσβαση σε δεδομένα ως προς τις ροές της ηλεκτρικής ενέργειας σήμερα, γιατί κάθε, σύστημα, κάθε διαχειριστής μάλλον συστήματος ε, ε, διανομής ε, παρακρατάει τα δεδομένα αυτά και δεν τα δίνει. Έτσι λοιπόν, τουλάχιστον σε περιφερειακό επίπεδο, θα ήταν καλό να έχουμε ένα συντονισμό, ένα καλύτερο συντονισμό μεταξύ των διαχειριστών συστημάτων διανομής, ε, τον, τα δεδομένα λοιπόν όλα αυτά, τα οποία θα μας επέτρεπαν να έχουμε πιο πολλά δεδομένα, πιο πολλές πληροφορίες και ως εκ τούτου μια καλύτερη βάση σχεδιασμού. Και άλλες πτυχές, μια άλλη καλύτερα πτυχή που θα ήθελα να υπογραμμίσω, γιατί πριν από μερικούς μήνες ε, με είχε απασχολήσει το πρόγραμμα «Ήλιος», με βασική ιδέα στην Ελλάδα ε, και χάρη σε γερμανικά ε, κονδύλια να κατασκευαστούν μεγάλης κλίμακας ε, φωτοβολταϊκές μονάδες. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω όμως είναι πώς είναι δυνατόν τα φωτοβολταϊκά τη σήμερα ημέρα να είναι ως επένδυση πιο ε, αποδοτική, πιο φθηνή στη Βαβαρία από ό,τι στην Ελλάδα. Το ξαναλέω, πιο φθηνό στη Βαβαρία παρά στην Ελλάδα να κατασταθούν φωτοβολταϊκά. Ωστόσο, ωστόσο, πριν θεωρήσετε ότι είμαι ανόητος, θα ήθελα να σας επισημάνω ότι η απόκληση που έχουμε ως προς την ε, ε, ηλιακή ενέργεια, την ηλιακή ε, ακτινοβολία, είναι πολύ χαμηλότερη από την απόκληση που υπάρχει ως προς το κόστος της επένδυσης. Γι' αυτό η Ελλάδα είναι πολύ πιο ακριβή σαν επένδυση στα φωτοβολταϊκά. Και γι' αυτό θα πρέπει να κοιτάξουμε την διάσταση των απευθεία επενδύσεων. Είναι πολύ πιο ακριβό αυτή τη στιγμή στην Ιρλανδία να γίνουν επενδύσεις δικτύου ε, διότι παρεμβαίνει ο κρατικός παράγοντας, ο κρατικό τομέα. Λοιπόν, ίσω θα έπρεπε να δώσουν περισσότερη έμφαση στις ε, πρωτοβουλίες Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να μειώσουν το κεφαλουχικό κόστος, ιδιαίτερα για τις χώρες οι οποίες σήμερα έχουν πολύ ψηλό κεφαλουχικό κόστος να ε, πληρώσουν. Ο κύριος Κοσέ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ε, δεν άκουσα από τους δύο εισηγητές ε, της εκθέσεως κουβέντα για το μέγεθος των μέσων παραγωγής ως προς την ε, τις ανανεώσιμες πηγές και την αναλογία ως προς την τοπολογία στα ευρωπαϊκά δίκτυα. Πλην όμως υπάρχει μια σαφής αναλογία. Εάν δηλαδή θεωρεί κανείς ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να απορρεύσουν από μεγάλα κέντρα παραγωγής, δηλαδή από κάποιες κεντρικές μονάδες, θα πρέπει να στραφούμε στα ε, δίκτυα υψηλή τάσεω και ούτω καθεξή. Αν όμω, αντίστροφα, βάζει και τον όσο λέει ο αγαπητό φίλο Ρίφκιν στο βιβλίο του, θεωρήσουμε ότι κάθε σπίτι, ε, κτίριο, οικοδομικό τετράγωνο, ακόμη και ηλεκτρικό αυτοκίνητο μπορεί να αποτελέσει πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Δηλαδή έχουμε εκατομμύρια μικρών, μικρής κλίμακας πηγών ηλεκτρικής ενέργειας. Στην περίπτωση αυτή το δίκτυο το ίδιο δεν έχει καθόλου την ίδια μορφολογία, τοπολογική διαμόρφωση ε, με αυτή των μεγάλων κεντρικών ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων. Τι βλέπετε λοιπόν εσείς ως όραμα το 2050. Και δεν μιλάω για πηγές παραγωγής. Κοιτάξτε, μικρές μονάδες, πάρα πολύ αποκεντρωμένες, πάρα πολύ ε, διάσπαρτες, μεν ή ε, μόνο μεγάλες κεντρικές ε, μονάδες δε, γιατί αλλάζουν τα πάντα ανάλογα με το τι θα... Ε, τι εξέλιξη έχουμε. Επίσης κάτι άλλο, και το λέω καθώς ήμουν πρώην βουλευτή στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, οι ροέ αλλάζουν επίση και κάποιο ε, παλιό συνάδελφο βουλευτή από την Γαλλική Εθνοσυνέλευση έλεγε ότι φτάνει πια αυτό η ιστορία με τα δίκτυα, διότι ούτω ή άλλω δεν μπορούμε να τηρήσουμε την, ε, τους νόμους του Κίρσοφ και ω εκ τούτου θα πρέπει να ψηφίσουμε καινούριου. Ευχαριστώ πολύ. να ακούσουμε ακόμη έναν συνάδελφο, μία συνάδελφο και να δώσουμε το λόγο μετά στους ομιλητές μας. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πολύ σημαντική και απαραίτητη ε, νομοθεσία και το ε, βλέμμα προς το μέλλον που μας προσφέρατε ήδη βλέπουμε ότι υπάρχει δυνατότητα να υλοποιηθούν τα πάντα. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε στο 2040. Έτσι λοιπόν, εμπόδια είναι ουσιαστικά τα κοινωνικά. Τι αυτά. Πώς λοιπόν θα μπορούσαμε με καλύτερες πολιτικές επιλογές να πείσουμε τον κόσμο ότι μπορούν να, μπορεί να εξασφαλίσει έναν πλανήτη πιο καθαρό, πιο υγιή, χάρη στις ανανεώσιμες πηγές. Ώστε να πει και ότι μπορεί χάρη σε αυτές τις νέες δυνατότητες να εξασφαλίσει και περισσότερες εργασίες. Διότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προσφέρουν δυναμικό για νέες θέσεις εργασίας και προοπτική για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακαλώ το λόγο ουχή. Και ως εκ τούτου δίνω το λόγο για να απαντήσουν σε ερωτήσεις τους δύο οι συγητές των, της εκθέσεως με τη σειρά. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις σας. Λογικό είναι να προσπαθήσουμε βέβαια να απαντήσουμε τις ερωτήσεις που μας κάνατε και όσες άλλες βρήκαμε. Αν μιλάμε για ενσωμάτωση ε, ανανεώσιμων, αυτό το οποίο έχουμε είναι μια πάρα πολύ μακροσκελή εξίσου με πάρα πολλές μεταβλητές και το ζήτημα βεβαίως που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι να προσπαθήσουμε να βρούμε τη σωστή λύση και όλες αυτές οι μεταβλητές είναι εξίσου σημαντικές. Σημαντικό είναι να υπογραμμίσουμε τη σύσταση που κάνουμε για περισσότερη έρευνα και επιστημονική συζήτηση στον τομέα αυτών και αυτό είναι βασικό κομμάτι της μελέτης, σας, μας. Να τονίσω κάτι για τα διάφορα, τα διάφορα εμπόδια, αν μπορούν να εμποδίσουν τις αγορές. Ε, είναι ε, λοιπόν σημαντικό ερώτημα. Εάν ε, τα εμπόδια αυτά τα οποία βρήκαμε μπορούν να τροχοπεδίσουν την κατάσταση. Υπάρχουν λύσεις, ε, αλλά βεβαίως θα απαιτηθεί πολιτική βούληση και έρευνα και βεβαίως αφοσίωση για να δώσουμε μια συνέχεια. Και οπωσδήποτε η κοινωνική αποδοχή είναι πάρα πολύ σημαντική αν μπορούμε να εξηγήσουμε τα ωφέλη του συστήματος αυτούς τους κοινωνικούς μας εταίρους θα είναι νομίζω στο πλευρό των νέων εξελίξεων. Θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον Ματίας για τις υπόλοιπες ερωτήσεις. Well, I'll, try to answer um, main groups of Τις βασικές ερωτήσεις, μία για την αποθήκευση, μία για τις επενδύσεις στα δίκτυα και ένα άλλο για τις ίδιες τις ανανεώσιμες. Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Ένα ερώτημα ήταν πώς θα έπρεπε να κοιτάξουμε τα απόβλητα ως κάτι το ανανεώσιμο. Στατιστικά νομίζω ένα 40% θεωρείται ανανεώσιμο και ένα 60% είναι ορυκτό, αλλά είναι πολύ μικρό ποσοστό ακόμα και αν όλα τα οικιακά και λοιπά απορρίμματα πήγαιναν για παραγωγή ενέργειας θα ήταν ένα πολύ μικρό ποσοστό της κατανάλωσης της ενέργειας. Οπότε οι ανανεώσιμες πηγές, ε, οι άλλες ανανεώσιμες πηγές, είναι μάλλον οι σημαντικότερες ποσοτικά. Επίσης άλλο ερώτημα, πως θα έπρεπε να κοιτάξουμε και άλλες πηγές ενέργειας γιατί είναι πολύ φτηνότερες και τελικά ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό, ο καταναλωτής. Αν δείτε την εξέλιξη του κόστους, οι ανανεώσιμες ε, γίνονται φτηνότερες, αν δείτε τα φωτοβολταϊκά μιλάμε για διψήφια ποσοστά ετήσιας μείωσης του κόστους. Έχουμε ήδη φτάσει σε ένα επίπεδο που τα καθιστά ελκυστικά για νοικοκυριά και ε, έχουμε φτάσει πλέον σε ισότητα δικτύου, δηλαδή είναι φτηνότερο να παράγει κανείς σπίτι παρά να παίρνει από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό θα γίνει σε κάνα δύο χρόνια από σήμερα θα φτάσουμε εκεί. Οπότε θα έλεγα πως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν το κόστος μέσω μακροπρόθεσμα τώρα. Να έρθουμε στο ερώτημα των επενδύσεων στα δίκτυα. Τονίσαμε στην ανάλυση μας ε, και στην παρουσίασή μας πως ε, η άποψη από πάνω προς τα κάτω είναι σημαντική αλλά πάντα με μια αίρεση στην ανάλυση μας. Η ανάλυση μας δεν συμπεριλαμβάνει το πακέτο υποδομών, γιατί εμάς η ανάλυση μας ολοκληρώθηκε μέσα Οκτωβρίου, ακριβώς πριν προταθεί από την Κομισιόν το πακέτο αυτό. Οπότε είναι σημαντικό, πρέπει να δούμε από κοντά το τι προτείνει το πακέτο. Αυτό το οποίο βλέπουμε λοιπόν, και αυτό δεν βασίζεται σε λεπτομερή ανάλυση, είναι πως δεν υπάρχει αρκετή τέτοια προσέγγιση ε, από πάνω προς τα κάτω στους κανονισμούς που προτείνονται αυτή τη στιγμή. Τελευταία ερώτηση αφορούσε την αποθήκευση, εάν ε, είναι το αποπέδι θα έλεγε κανείς ή μια δευτερεύουσα προτεραιότητα της επέκτασης του δικτύου. Ναι, πράγματι στις περισσότερες περιπτώσεις θα είναι φτηνότερη η επέκταση του δικτύου, αλλά και η αποθήκευση μπορεί να είναι γρηγορότερη και ίσως φθηνότερη κατά τόπους. Ειδικά στο δίκτυο διανομής ε, είναι η πιο ενδιαφέρουσα οικονομικά περίπτωση, η αποθήκευση, να αντικαταστήσουμε την ε, επέκταση του δικτύου που διαφορετικά θα ήταν απαραίτητη και μιλάμε για μέσο πρόθεσμα σε 5-10 χρόνια. Οπότε στο τοπικό επίπεδο είναι μια ενδιαφέρουσα επιλογή. Τώρα... Για μεγάλης ε, κλίμακος συστήματα τα οποία θα έχουν εποχιακή αποθήκευση ε, ενέργειας. Ο κύριος Πόντι αναφέρθηκε στο υδρογόνο ως μια βασική μορφή ε, αποθήκευση του ηλεκτρισμού. Μόνο με χημική μορφή μπορεί να αποθηκευτεί σε μεγάλη κλίμακα ο ηλεκτρισμός, είτε ως υδρογόνο ή ή ως συνθετικό φυσικό αέριο που παράγεται με τον ηλεκτρισμό. Είναι θέμα λοιπόν η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο απαιτεί την πιο έντονη ανάπτυξη τεχνολογιών από όλες τις τεχνολογίες τις οποίες αναφέραμε σήμερα, αλλά ιδίω σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρισμό, σημαίνει ότι έχει και κάποια μειονεκτήματα, κυρίως το κόστος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, σας ευχαριστούμε και τους δύο εισηγητέ, δύο παρουσιαστέ τη έκθεση αυτή και μπορούμε να προχωρήσουμε στι ψηφοφορίε. Κυρία Πρόεδρε, έχω να σας θέσω ένα ερώτημα. Εγώ έχω συζητήσει σε όλες αυτές τις συζητήσεις και σας ευχαριστώ για την ενημέρωση που πήρα. Αλλά το έγγραφο αυτό, το οποίο μας έχει διανεμηθεί, αν είναι διαθέσιμο στη μητρική γλώσσα των βουλευτών θα ήθελα να ξέρω. Le peuple. Σίγουρα θα μεταφραστεί σε όλες τις ε, γλώσσες, αλλά αυτή τη στιγμή δεν ήταν διαθέσιμο. Περνάμε λοιπόν στη ψηφοφορία όπως σας έλεγα. Έχουμε την έκθεση Τσίτσεστερ για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο, για τον Ευρωπαϊκό Φορέα Ασφάλειας των Δικτύων, την ΕΝΙΣΑ. Πριν αρχίσουμε την ψηφοφορία, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι όταν φτάσουμε στον κατάλογο ψηφοφορία στο σημείο της φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και του ηλεκτρισμού, στο, στην 102, 103, 104. Ήθελα να ζητήσω να ψηφιστούν 103 και 104 ως προσθήκες στην 102, όχι χωριστά. Η 103 και 102 φορολόγηση ενεργειακών προϊόντων ως προστίκες στην 102. Όταν φτάσουμε στο σημείο αυτό, λέει η πρόεδρος. Ψηφίζουμε λοιπόν. Συμβαστική τροπολογία 1. <clears throat> Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται άρθρο παράγραφος 4 τροπολογία 57 τσίτσεστερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 3 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Άρθ, τροπολογία, παράγραφος 6, τροπολογία 210, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άρθρο 7, παράγραφος 1, τροπολογία 74, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 25 λίμπε, ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 213 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 75 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 214 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 77 σε δύο, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 215 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 78 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 94 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 95 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 97 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται.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 κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6. Παρακαλώ διαδικαστικά κυρία Ένιγκ. Κυρία Πρόεδρε, για την τροπολογία συμβασμού 6 θέλουμε μία διαφοροποιημένη ψηφοφορία για το να είναι η έδρα της ε, Υπηρεσία στην Ελλάδα, αλλά να είναι το κέντρο της στην Αθήνα. να χωρίσουμε την δεύτερη γραμμή της τροπολογίας από την πρώτη. Γιατί αν υπάρχει η δέσμευση να έχουμε αυτή την υπηρεσία στην Κρήτη, δεν μου φαίνεται σωστό να είναι η υπηρεσία στην Κρήτη και ένα μέρος του προσωπικού της, της γραμματείας της ή οτιδήποτε να είναι στην Αθήνα. Γι' αυτό ζητώ μια διαφοροποίηση στην ψηφοφορία δεν μπορώ να δεχτώ ε, χωριστές ε, ψηφοφορίες σε μια συμβαστική τροπολογία, λέει η Πρόεδρος. Δεν γίνεται αυτό, δεν επιτρέπεται. Θα έπρεπε να το είχατε ζητήσει εκ των προτέρων. Συμβαστική 6 λοιπόν, ψήφι υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 115 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ λίμπε κατά αποχές εγκρίνεται. 237 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 239 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7α. Σε 7α ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Θα κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία. 7α. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 7β. Ψήφι πέρα κατά άποχες εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 126. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 127. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 128. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 131. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 135. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 11. Υπέρ. Όχι. Όχι. Όχι. Πηγαίνουμε. Ναι. Συγγνώμη, συγγνώμη. Είχε ακυρωθεί. 17 Τσίτσεστερ ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 11 Λίμπε υπέρ. Λίμπε 11 στην αιτιολογική σκέψη 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Υπαριθμόν 23 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 150 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 8, όχι, όχι με συγχωρείτε. 26 27 λέει πρόεδρος. Κατά αποχές εγκρίνεται. 8 κατά αποχές εγκρίνεται. 153 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίσαμε την 26 καθώς και την 151 που ταυτίζονται. Τις ψηφίσαμε από κοινού. Εντάξει λέει. Εντάξει. Και τώρα που είμαστε. 154 και 155 σε δύο τμήματα. Ταυτίζονται δύο τροπολογίες. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ψήφι Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα. 30. <clears throat> Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 156. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 124 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 125 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κύριε Πρόεδρε, η 125 εκπίπτει. Όχι, όχι, συγγνώμη. Συγγνώμη, συγγνώμη. Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τελική ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Πέρας. Μια στιγμή ακόμα. Πέρας. Ωραία. 51 ψήφοι υπέρ, 3 κατά και 52 μάλλον, 52 γιατί ήταν χωρίς ε, κάρτα. 52 υπέρ, 3 κατά και μία αποχή. Θαύμαση. Συγχαρητήρια κυρία Τσίτσεστερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους ε, συναδέλφους ε, για την ψηφοφορία και είμαι ικανοποιημένο από το αποτέλεσμα. όμω, ζητώ να αναβάλουμε την ψηφοφορία επί του νομοθετικού ψηφίσματος για να έχουμε περισσότερο χρόνο να συζητήσουμε με το Συμβούλιο και την Κομισιόν. Θα ήθελα να αναβληθεί λοιπόν η ψηφοφορία επί του νομοθετικού ψηφίσματο. Bene, abbiamo terminato. Passiamo Έχουμε κλείσει, εντάξει. Πάμε στην επόμενη έκθεση. Συμφωνείτε όλοι. Το νομοθετικό ψήφισμα θα αναβληθεί η ψήφισή του. Γραμματεία λέει όχι. Δεν έχει νόημα το ψηφίσουμε. Αφήνουμε λοιπόν το νομοθετικό ψήφισμα και ερχόμαστε στη δεύτερη, στη δεύτερη ψηφοφορία. 6. Έκτο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον και καθορισμός προτεραιοτήτων για το 7ο πρόγραμμα δράσης υπέρ του περιβάλλοντος. Η συγγήτρια είναι η κυρία Κριστίνα Γκουτιέρες Κορτίνες, τροπολογία 1, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ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 αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ. Θέλετε έλεγχο για την 17. Ε, Έλεγχος ηλεκτρονικός για την 17. Πέρας. Απορρίπτεται.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 κατά αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 32, συγγνώμη, συγγνώμη, εγκρίνεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 33 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έλεγχος στην 33.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 Ήταν 38 αυτή λοιπόν. Πάμε στην 39, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 40 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 41 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 42 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται τελική ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Πέρας. 51 υπέρ, καμία ψήφος κατά. 52 υπέρ, ναι, καμία κατά. Τέσσερις αποχές. Περνάμε στο επόμενο σημείο. εξασφάλιση της ζωής, φυσικό κεφάλαιο, στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την βιοπικιλότητα για το 2020. Συμβαστική τροπολογία Α. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Β, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, 6, τροπολογία 6, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική γάμα σ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική ε, τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική D δέλτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 20 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 22 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 23 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 24 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 25 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται να ελέγξουμε την 30 επαλήθευση Πέρα τη ψηφοφορία. 41 κατά, 14 πέρ. Είναι προφανέ ότι απορρίπτεται. Και ευχαριστώ 29 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 31 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και τελική ψηφοφορία με ονομαστική κλείσει. Παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Πολύ καλά, 54 υπέρ, μία ψήφος αποχής. Και τώρα παρακαλώ να περάσουμε στο θέμα των τροφών για βρέφη και μικρά παιδιά. Παρακαλώ. Ε, χαίρετε. Εκ μέρου του κυρίου Τάκουλα, του εισηγητού, θα ήθελα να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις, λέει ο κύριος Ρόντα, για την υπόθεση αυτή. Σε συμφωνία με τους κοιόδης εισηγητέ των λοιπόν ομάδων έχουμε κατά μνήμη τις ε, σε δύο βασικές ε, ομάδες, α που αφορά το γάλα για τα μικρά παιδιά και β για την κατηγορία εκείνων που έχουν δυσανεξία στην ε, Θεωρούμε ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντο αρμόδια για τη δημόσια υγεία θα ήταν καταλληλότερη να ψηφίσει το θέμα αυτό και γι' αυτό προτείνουμε να απορριφθούν αυτέ οι τροπολογίε για να εισαχθούν στη συνέχεια στο επεξηγηματικό υπόμνημα τη ε, γνωμοδότηση που θα εξηγεί τι πτυχέ αυτέ, τα δεδομένα αυτά και θα ζητεί από την Επιτροπή Περιβάλλοντο και Δημόσια Υγεία να αναλύσει την κατάσταση και τι τροπολογίε αυτέ ει βάθο. Ευχαριστώ θερμά. Καλώς, ευχαριστώ κύριε Ρόντε. Άρα θα ακολουθήσουμε αυτή την πρόταση και προχωρούμε με την υπαριθμόν 53. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Να επαληθεύσουμε. 56. Πέρασε. 34 υπέρ 18 κατά. Εγκρίνεται. 57 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. Υπαριθμών 4 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 59 σε 4 τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τέταρτο τμήμα. Καλώς. Ε, έληξε το απερίφθιο ολόκληρο. Τώρα 60 τώρα παρακαλώ υπέρ. Κατά. Υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία παριθμών 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το 63 τώρα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 6, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 64, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 66 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. Εγκρίνεται διορθώνει ο πρόεδρος. 67 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 73 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 87 καταπίπτει, 89 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 92 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 1 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 22, τρία τμήματα, τέσσερα τμήματα, διορθώνει ο Πρόεδρος, πρώτο τμήμα παρακαλώ υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται και καταπίπτουν τα υπόλοιπα τρία. Περνάμε τώρα στη συνανθρωπολογία 23 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 24 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ. Θα επαληθεύουμε την 24. 24 επαληθεύσει άρχεται η ψηφοφορία. 28 υπέρ. 25 κατά. Εγκρίνεται. Η 24. Στη, εκεί στις προφορές 25 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 31 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 34 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 35 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 36 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και ομού σε δύο ομάδες όπως είπαμε. Πρώτη ομάδα υπέρ, κατά. Δεν το βλέπω ξεκάθαρα, ας επαληθεύσουμε για, το πρώτο, για την πρώτη ομάδα τροπολογιών. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Πέρασε ψηφοφορίες, 28 υπέρ, 27 κατά. Σωστά αφέβαλα. Εγκρίνεται πάντως. Δεύτερη ομάδα. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Να επαληθεύσουμε την ψηφοφορία για το Β, για τη δεύτερη ομάδα. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία για τη δεύτερη ομάδα. Πέρας ψηφοφορία για τη δεύτερη ομάδα. 22 υπέρ, 33 κατά και ως εκ τούτου απερίφθη. Τώρα έχουμε την υπαριθμόν 7 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απεριφ... Τελική ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Πέρας. 42 υπέρ, 11 κατά, μία αποχή εγκρίνεται. Και τελευταία ψηφορία. Τροποποίηση της οδηγίας του Συμβουλίου σε σχέση με το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη φορολογία ενεργειακών προϊόντων και ηλεκτρισμού. Η κυρία Ούλσκοκ θέλει να κάνει κάποια παρατήρηση. Όχι. Εντάξει. Βεβαίως θέλω να πω κάτι. Σε σχέση με την τροπολογία Πού να είμαστε τώρα. 103 και 104 να θεωρηθούν ότι είναι προστίκες να μην εκπέσουν όπως ε, λανθασμένα αναφέρεται στον κατάλογο ψηφοφορίας, να ψηφιστούν ως προσθήκες. Ωραία, ωραία. Ναι, ναι, το έχουμε ήδη δει αυτό. Λοιπόν, τροπολογία 43, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ. Όχι, όχι, όχι, όχι, βλακίες. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίντ, 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίντ, 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 <clears throat> υπέρ έλεγχος για την 53 βεβαίως άρχεται πέρας είχατε δίκιο 25 υπέρ 30 κατά απορρίπτεται. 53 απορρίπτεται λοιπόν. Απερίφθη 53. 54 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Check, check. Άρχεται η ψηφοφορία. Για την 54. Πέρας. 34-21 εγκρίνεται πράγματι. «55 και 56 ταυτίζονται. Ψηφίζουμε μαζί. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 5 παρακαλώ. Έλεγχος για την 55 και την 56 βέβαια. Πέρας. 34 υπέρ, 20 κατά, όπως και πριν. «55 και 56 μαζί» λέει η πρόεδρος. Κατά. Α, αφού τις ψήφισαν προηγουμένως. Συγγνώμη. 5. 5. 5 και 60. Που είναι μαζί. Υπέρ κατά αποχές υπάρχει κάποια αμφιβολία. Δεν ξέρω αν σηκώνετε όλοι τα χέρια σας ή όχι, ας κάνουμε ένα έλεγχο. Πέρας. 34 υπέρ 19 κατά. Λίγα χέρια σηκώθηκαν και δεν ήταν σαφές το αποτέλεσμα. 61. <clears throat> Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6 και 62 που είναι ταυτόσιμες. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 7 και 64 που ταυτίζονται και πάλι υπέρ. Κατά αποχές εκδίδονται. 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 73 λέει η πρόεδρος. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ναι, έπρεπε να ψηφίσουμε και την 72 λέει η πρόεδρος γιατί δεν απερίφθη, δεν εγκρίθηκε η 72 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 79 <clears throat> υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 83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 90 και 91 είναι ταυτόσιμες υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. Θέλετε έλεγχο. 90 και 91, ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρας. Είκοσι υπέρ, 34 κατά. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 93 κατά αποχές εγκρίνεται 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 96 και 97 είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 100 σε δύο τμήματα. Τμήμα 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 105 λέει η πρόεδρος κατά αποχές απορρίπτεται. 106 παρακαλώ παρακαλώ. Συγγνώμη κυρία Πρόεδρε, όπως είχε ζητήσει η κυρία Ουλσκοκ προηγουμένως, είπατε ναι, να ψηφίσετε 103-104 ως ε, προσθήκη. Ναι, ναι, συγγνώμη, το ξέχασα λέει η πρόεδρος. 103 και 104 θα τις ψηφίσουμε. Σαν προσθήκη στην 102. Η 103 προσθήκη στη 2 και η 104 στην 3. 103. Σαν προσθήκη στην 102. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται η 104 δεν έχει νόημα πια. Αν να ψηφίσουμε και την 104 σαν προσθήκη υπέρ, κατά απορρίπτεται ούτως ή άλλως. Έλεγχος. 28 υπέρ, 25 κατά. Επομένως εγκρίνεται. που λέει η γραμματεία ότι είχαμε ξεχάσει να ψηφίσουμε την 92. Συγγνώμη, πρέπει να ψηφίσουμε την 92 γιατί οι 90 και 91 δεν είχαν εγκριθεί. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 105. Έλεγχος για την 92, βεβαίως. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 105. 105. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 108. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 109 υπέρ. Συγγνώμη, την 107 την ξεχάσαμε. 107 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 108 την ψηφίσαμε. 108 ονομαστική κλίση λέει η πρόεδρος. Δεν την ψηφίσαμε ονομαστική κλίση. Άρχεται. Όχι, όχι, ηλεκτρονικό έλεγχο κάνουμε στην 108. Υπήρχε αίτηση για, για έλεγχο. Πέρας. 29 υπέρ 24 κατά γίνεται δεκτή. 109 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 110 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 111 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 112 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 113 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ένα, ένα, τέσσερα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αιτιολογικές σκέψεις, 13, υπέρ, Έλεγχος ηλεκτρονικός είναι 114. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 32 υπέρ 22 κατά εγκρίνεται. Ωραία. 110, τροπολογία 13, συγγνώμη, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2 και οι 20 είναι ταυτόσιμες. Ψηφίσουμε. Ψήφι Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Έλεγχος για τη δύο και η Πέρας. 29-24 εγκρίνονται.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 Έλεγχος για 32. Άρχεται. Πέρας. Το ΕΛΚ έχει ένα παραπάνω, βγαίνω τον... βγάζω τον εαυτό μου εγώ. Πέρας ψηφοφορίας. 26 υπέρ, 25 κατά, εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος. Ψηφίζουμε. Άρχεται. Πέρας. Πέρας. 26-26 ισοψηφία απορρίπτεται. Απορρίπτεται. «35» λέει πρόεδρος υπέρ, κατά, απόχες, απορρίπτεται. 36 υπέρ, κατά, απόχες, απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά, απόχες, απορρίπτεται. Έλεγχος. Έλεγχος για την τρία. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 38 υπέρ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 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, τελική, τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας. Μια στιγμή, λέει πρόεδρος. Πέρας ψηφοφορία. ...27 υπέρ, 28, 25 κατά με δύο αποχές, γίνεται δεκτή, 27-25. Πέρας της περίοδου ψηφοφοριών, αν θέλετε λοιπόν να ξεμουδιάσετε και μετά περάσουμε στις δύο τελευταίες εκθέσεις.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 Bene, allora passiamo al punto numero 10 dell'ordine del giorno. Σημείο 10 της ημερησίας διάταξης. Μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών σε διακυβερνητικέ συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της ενέργειας. Βλέπετε να κρατήσει 45 λεπτά αυτή τη συζήτηση. 112 τροπολογίες έχουν παρουσιαστεί. Οι περισσότερες στα αγγλικά, αλλά υπάρχουν οι μεταφράσεις τους. Και έχουμε κάνει μια πρώτη συζήτηση στην προηγούμενη συνεδρίασή μας. Θα δώσω το λόγο στην κυρία, στον κύριο Κάρινς για τις κατατεθήσεις τροπολογίες. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Ε, θέλω να ακούσω τι έχουν να πούν και οι συνάδελφοι. Πρώτα απ' όλα να πω ευχαριστώ πολύ ε, όσους υπέβαλαν τροπολογίες, κάποιες ήταν ενδιαφέρουσες, κάποιες άλλες μου προξένησαν απορία το βασικό πράγμα που θα ήθελα να πω. Εγώ θεωρώ το νομοθέτημα αυτό πολύ σημαντικό και πρέπει να περάσει γιατί θεωρώ πως χρειαζόμαστε στην Ευρώπη ε, η Κομισιόν να έχει ένα ρόλο να εμπλέκεται σε διακυβερνητικές συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και παρόχων ενέργειας από τρίτες χώρες ε, να είναι αυτές οι συμφωνίες σύμφωνες με το κοινοτικό δίκαιο που είναι ο κύριος στόχος και δευτερεύον στόχος είναι η Ευρώπη να δημιουργήσει μια κοινή φωνή, μια κοινή προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις ε, προμήθειας ενέργειας για να ωφεληθούν όλοι οι καταναλωτές της Ένωσης. Μου φαίνεται πως είναι σαφές πως θα έχουμε κάποια αντίσταση από αρκετά κράτη-μέλη ε, επί του νομοθετήματος ε, στο σύνολό του, ειδικά οποιαδήποτε πτυχή ε, θα είναι υποχρεωτική. Γι' αυτό θεωρώ πως είναι ιδιαίτερα σημαντικός κοινοβούλιο να έχουμε όσο το δυνατόν πιο ενωμένη στάση για να μπορούμε να ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση στις συζητήσεις με το Συμβούλιο και την Κομισιόν. Έχω δύο σχόλια τώρα, ένα από τα οποία είναι μία ερώτηση για τις ε, υποβληθήσεις τροπολογίες. Το πρώτο είναι η φύση των εμπορικών συμφωνιών. Αν διαβάσει κανείς τις διάφορες τροπολογίες βλέπει πως έχουμε δύο, τις δύο πλευρές θα έλεγε κανείς της συζήτησης. Κάποιες λένε πως καμία εμπορική συμφωνία δεν πρέπει να συμπεριληφθεί κατά τρόπο ακόμα και αν είναι διακυβερνητικές από την άλλη έχουμε τροπολογίε που λένε όχι μόνο οι διακυβερνητικέ συμφωνίε πρέπει να καλύπτονται, αλλά και όλες οι εμπορικέ. Αυτό το οποίο προτείνω είναι κάτι στη μέση. Να κρατήσουμε δηλαδή το σκεπτικό εδώ πέρα της νομοθεσίας, ε, όπως το πρότεινε η Κομισιόν, δηλαδή η νομοθεσία που θα καλύπτει διακυβερνητικές συμφωνίες, αλλά και τις πτυχές εκείνες των εμπορικών συμφωνιών που αναφέρονται ρητός στις διακυβερνητικές συμφωνίες και αυτές θα υποβάλλονται στην Κομισιόν. Και στο άρθρο 7, νομίζω, είναι το άρθρο που αφορά την εμπιστευτικότητα και είναι εξαιρετικά σημαντικό να συμπεριλάβουμε στην νομοθεσία διατύπωση που θα λέει πως όταν τμήματα της συμφωνίας υποβάλλονται στην Κομισιόν για αξιολόγηση να παραμείνουν εμπιστευτικά και να μην ε, μεταδοθούν σε άλλα κράτη μέλη. Οπότε μόνο η Κομισιόν θα εξετάζει την νομιμότητα ή το συμβατό με το κοινοτικό δίκαιο. Αλλά οπωσδήποτε οι εμπορικές πτυχές δεν θα ε, κοινοποιηθούν στα άλλα κράτη-μέλη. Αυτή είναι η ε, παράκλησή μου προς τις δύο πλευρές. Το δεύτερο θέμα το οποίο θα ήθελα να θίξω είναι στις τροπολογίες 112, 114 και 16 για τη συμπερίληψη ή μη ε, μιας ε, αναφοράς σε επενδυτικές συμφωνίες. Εάν διαβάσει κανείς την ομοθεσία και τις τροπολογίες που εγώ τις διάβασα, απόρρισα για το, και δεν είμαι σίγουρος για το εάν είναι σωστή αυτή η ιδέα και για το εάν κολλάει εδώ πέρα. Και διαβουλεύτηκα και με την Κομισιόν και η Κομισιόν, ε, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, δεν αντιλαμβάνεται γιατί ακριβώς πρέπει να συμπεριληφθούν επενδυτικέ συμφωνίες σε αυτήν εδώ την νομοθεσία. Η Κομισιόν λέει πως καλύπτονται από άλλη νομοθεσία. Οπότε αυτό είναι το ερώτημά μου προς τους συναδέλφους που συνέταξαν αυτές τις τροπολογίες. Ποιο είναι το επιχείρημα εδώ πέρα. Δεν είναι κακό, αλλά έτσι, για λόγους ε, κομψότητας ε, δεν βλέπω εγώ πώς ταιριάζει εδώ πέρα. Να σημειώσουμε επίσης, αύριο θα συναντηθώ με τους κοιόδης εισηγητές των άλλων ομάδων για να συζητήσουμε αρκετές συμβιβαστικές τροπολογίες που συντάσσω αυτή τη στιγμή. Ε, όσον αφορά τα ζητήματα του χρονοδιαγράμματος, έχω μία πρόταση η οποία βεβαίως είναι κάπου στη μέση. Η Κομισιόν λοιπόν μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά και να μην υποφέρει και ο κλάδος άδικα. Μπορώ να σχολιάσω διάφορα ζητήματα, αλλά αυτές είναι οι δύο πτυχές που θα ήθελα εγώ να θίξω, οι εμπορικέ συμφωνίες και η πρότασή μου, δηλαδή να ακολουθήσουμε μία μέση οδό και το ερώτημα προς συναδέλφους που έχουν καταθέσει τροπολογίες για τις εμπορικές ε, συμφωνίες. Δεν βλέπω το λόγο η Κομισιόν τουλάχιστον ε, στη συζήτηση μαζί μου δεν είχε κάποια επιχειρήματα. Δεν ξέρω, ε, ίσως οι συνάδελφοι μπορούν να με πείσουν, ε, είμαι ανοιχτό. Θα μείνω σε αυτά και θέλω να ακούσω και τους συναδέλφους. Ευχαριστούμε κύριε Κάρενς. Κύριος Λάγκα. Σκιώδης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ καταρχάς τον εισηγητή. Έχετε νομίζω ακολουθήσει στην ορθή στάση, αναζήτηση δηλαδή συμβαστική λύση. Το λέω αυτό διότι πιστεύω ότι είναι στι μεγάλη πρόκληση στην πραγμάτευση με το Συμβούλιο και γνωρίζουμε ότι στο Συμβούλιο πολλά είναι τα κράτη-μέλη τα οποία απορρίπτουν ε, αυτή την πρόταση, χρειάζεται πιστεύω συνένεση μεταξύ των πολιτικών ομάδων για να μπορέσουμε να σχηματίσουμε ένα ισχυρό μέτωπο έναντι του Συμβουλίου. Και είναι πολύ σημαντικό πιστεύω να δρομολογηθεί αυτό το νομοθέτημα, καθώς οι προκλήσεις της συναντιακής πολιτικής του μέλλοντος θα εξαρτηθούν προφανώς στην υλοποίησή τους και από τις σχέσεις με τα γειτονικά κράτη. Και έτσι όταν προσδιορίζουμε την πολιτική μας για το μέλλον θα πρέπει να γνωρίζουμε και τι είδους συμβάσεις μπορούν να επηρεάσουν αυτή την ενεργειακή πολιτική. Χρειάζεται λοιπόν συνένεση όπως έλεγα για να περάσει αυτό. Επίσης, κατά πρώτον πρόκειται για συμβάσει μεταξύ κρατών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ω εκ τούτου θεωρώ ότι δεν μπορούμε κάθε ε, τι να το υπαγάγουμε σε ιδιωτικού χαρακτήρα συμβάσεις, ε, ιδιωτικού δικαίου συμβάσεις. Άρα λοιπόν μιλούμε για διακρατικές συμβάσεις που αναπτύσσονται με βάση το διεθνές δίκαιο και αν ρητά προβλέπονται κάποια στοιχεία ιδιωτικού δικαίου, τότε τα κοιτάμε. Διαφορετικά στηριζόμαστε μόνο στο δημόσιο διεθνέ δίκαιο. Επίσης, συμμετοχή του Κοινοβουλίου αποτελεί φυσικά πολύ, σημαντικό, πολύ σημαντική πολιτική, διότι διαμορφώνουμε, εσύ διαμορφώνουμε την ενεργειακή πολιτική και ως εκ τούτου έχουμε δικαίωμα και να ενημερωνόμαστε ώστε να είμαστε βέβαιοι πως σε διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούμε να προσδιορίσουμε ένα κοινό δρόμο. Εδώ αυτό σημαίνει ταυτόχρονα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να επαληθεύει κατά πόσον αυτές οι συμβάσεις ε, έχουν θέση στη γενική ενεργειακή πολιτική και βέβαια την πολιτική για το κλίμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύω θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί περισσότερο από ό,τι μέχρι τώρα και δεν θα πρέπει να περιμένει απλώς μια πρωτοβουλία των κρατών μελών, θα πρέπει να αναλάβει τον συντονισμό και την επαλήθευση. Με τρόπο πιο αποφασιστικό. Και θα πρέπει ίσως να δούμε πώς μπορούμε να διατυπώσουμε το κείμενο έτσι να συμφωνήσουμε όλοι. Ε, για να προχωρήσω τώρα στη Συμφωνία Επενδύσεων. Στις Συμφωνίες Επενδύσεων υπάρχουν συμφωνίες οι οποίες συμπεριλαμβάνουν κάποια στοιχεία προστασίας των επενδύσεων όπως ο ενεργειακός χάρτης. Και εδώ θα ήθελα να το ενσωματώσουμε αυτό για να υπενθυμίσουμε στην Επιτροπή και Κύριο στο Συμβούλιο ότι όταν έχουμε να κάνουμε με τμήματα ε, του Συμφώνου Προστασία των Ενεργειακών Επενδύσεων σε μια σύμβαση, τότε και τα δικαιώματα και τα οι προνομίες του Κοινοβουλίου ως συνομοθέτη πρέπει να γίνονται σεβαστές. Και σε αυτό το βαθμό θα ήταν καλό να κάνουμε μια υπόμνηση και προς τους λοιπούς εταίρους μας ότι θα πρέπει ενδεχομένω να λαμβάνονται υπόψη και κάποιε άλλε διατάξει τη συνθήκη Λισαβόνα και ενδεχομένω να οργανωθεί διαφορετικά αυτό το σύνολο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρο. Σαντού. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Την προηγούμενη εβδομάδα στην Επιτροπή Εσωτερικού Εμπορίου ψηφίσαμε την ε, έκθεση, στηρίζεται, στηρίζουμε την πρόταση του κυρίου Καρίνς. Πριν μια εξαιρέσεω, την οποία δεν αντιληφθεί καλά. Την ε, απουσία βούλης από μέρους, ε, από πλευράς μελών της ΣΥΝΤΑ, ε, να τοποθετηθούν ω προ την ενεργειακή πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να την υποστηρίξουν. Ήδη νωρίτερα το απόγευμα συζητήσαμε τα ζητήματα των υποδομών και τις μεγάλες προκλήσεις προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Προφανώς τα όσα πράττουμε στο τομέα της ενέργειας σήμερα για να έχουν μια συνοχή και ενιαία προσέγγιση θα πρέπει να εγγράφονται στην ίδια δυναμική των μακροπρόθεσμων στόχων και έτσι και στη συζήτηση που θα έχουμε με τον κύριο Καρίνης αύριο θα ήθελα να επιμείνω ακριβώς στο σημείο αυτό που υπεγράμμισε και ο συνάδελφο ήδη, δηλαδή οτιδήποτε επένδυση γίνεται σήμερα στις συμβάσεις ε, που συνάπτουμε με τρίτα κράτη θα πρέπει να παρουσιάζει την ίδια συνοχή με τους κοινούς στόχους που έχουν προσδιοριστεί για το 2050 ή και ενωρίτερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ντελκαστείο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Γνωρίζουμε ήδη ότι αυτή η πρόταση της Κομισιόν είναι τμήμα μιας δέσμης που περιλαμβάνει αυτό το νομοθέτημα και μια ανακοίνωση η οποία θεσπίζει μια γενική στρατηγική για τις εξωτερικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θέματα της ενέργειας. Ευτυχώς είχαμε πολλές ευκαιρίες στο παρελθόν να συζητήσουμε αυτό το θέμα και στην Επιτροπή μας Και γι' αυτό θα σταθώ μονάχα σε ένα σημείο. και το οποίο είναι και αντικείμενο των λίγων τροπολογιών που εγώ κατέθεσα. Πρόκειται για την ε, διατύπωση αυτή, για τη ρήτρα που λέει ότι όλα αυτά τα οποία αποτελούν μια διακρατική συμφωνία μεταξύ ενός κράτους μέλους και ενός άλλου κράτους μέλους, σε όλες αυτές τις συμφωνίες να λαμβάνει κανείς με τον ίδιο τρόπο ακριβώς τις συμφωνίες μεταξύ εν, όπως λαμβάνει υπόψη συμφωνίες κράτους-κράτους διακρατικές, μια συμφωνία μεταξύ ενός κράτους και μιας κρατικής επιχείρησης ενέργειας. Όταν γίνεται λοιπόν συμφωνία μεταξύ ενός κράτους μέλους και μιας επιχείρησης που είναι δημόσιου χαρακτήρα, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση και το πλειοψηφικό κεφάλαιο, θα πρέπει να εφαρμόζονται όλοι οι μηχανισμοί διαφάνειας και πληροφόρησης, οι οποίες εφαρμόζονται και στις συμφωνίες καθαρά διακρατικού, διακυβερνητικού χαρακτήρα για, την, για, το περιεχόμενο αυτής της πρότασης. Δεν πρέπει κανείς να ξεχνάει ότι υπάρχουν επιχειρήσεις πολύ μεγάλης σημασίας που είναι δημόσιοι φορείς και στην περίπτωση αυτή όταν έρχονται σε συμφωνία με τρίτες χώρες παίζουν ένα καθοριστικό ρόλο αυτά. Ευχαριστώ, λέει η Ο κύριος Βιδάλ Κουάδρα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι στη φάση αυτή των συζητήσεων, στο στάδιο αυτό των συζητήσεων μάλλον, συμφωνούμε όλοι για την ανάγκη να υπάρξει ένας μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών σε σχέση με συμφωνίες οι οποίες έχουν διακυβερνητικό χαρακτήρα μεταξύ 100 μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών στον τομέα της ενέργειας. Και έχουμε όλοι μια συνένεση σε σχέση με τους λόγους που πρέπει να γίνεται κάτι τέτοιο, γιατί είμαστε μια ένωση η οποία βασίζεται στην αλληλεγγύη και είναι θεμητό ένα κράτος μέλος όταν συνάπτει μια συμφωνία με μια τρίτη χώρα μέσα στα πλαίσια της επιζήτησης του θεμητού κέρδους και των ωφελών στον τομέα της ενέργειας αυτό φυσικά μας χαροποιεί όλους, αλλά δεν θέλουμε μια τέτοια συμφωνία να θίξει άλλους εταίρους αλληλέγγυους άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί βρισκόμαστε μέσα στα πλαίσια μιας αλληλέγγυας ένωσης. Δεν θα είχε λοιπόν τότε νόημα να κάνει μια τέτοια συμφωνία. Συμφωνούμε λοιπόν σε νεολογικό και επίπεδο ιδεών. Τώρα όμως πρέπει να σταθούμε στα συγκεκριμένα θέματα. Πρέπει καταρχήν να δούμε ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής αυτής της συμφωνίας. Για ορισμένους συναδέλφους δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συμφωνίες μεταξύ ιδιωτικών φορέων. Για άλλους και εκεί Συμφωνική Κομισιόν μόνο αν υπάρχει μια συγκεκριμένη μνήα μέσα στην διακρατική συμφωνία θα πρέπει να ε, μα ενδιαφέρει αυτή η οδηγία και υπάρχουν άλλοι, μεταξύ των οποίων και η κυρία Δεκαστήλιο, η οποία προελάλησε, που θεωρούμε ότι όταν αυτή η διακυβερνητική συμφωνία είναι μεταξύ του κράτου και μια επιχείρηση δημόσιου χαρακτήρα μια τρίτη χώρα. τότε θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι δεν είναι μονάχα μια συμφωνία ιδιωτικού χαρακτήρα αλλά έχει και δημόσιες πτυχές. Μια συμβαστική πρόταση θα ήταν να κρατήσουμε την πρόταση της Κομισιόν και συγχρόνως να εξασφαλίσουμε ότι όλες οι πληροφορίες οι οποίες ε, είναι στα χέρια της Κομισιόν και θα ήθελε να τις ε, διαμοιραστεί με άλλα κράτη-μέλη, θα πρέπει να υπόκειται στη ρήτρα εμπιστευτικότητας. Αυτό νομίζω ότι είναι μια μορφή επίλυσης αυτών των προβλημάτων για τις σπάνιες περιπτώσεις, τις έκτακτες περιπτώσεις, όπου η εμπιστευτικότητα τρίτων εταιριών δύναται να θυγεί λόγω αυτής της συμφωνία. Μπορούν τα κράτη-μέλη τότε να πούν ότι αυτή η πληροφορία μπορεί να θεωρηθεί εμπιστευτική, ώστε η Κομισιόν να μπορεί να μην διαβιβάσει αυτή την πληροφορία στα άλλα κράτη-μέλη χωρίς να παραβιάσει το κείμενο τη οδηγία. Επίση, το θέμα τη συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις. Για ορισμένου. Είναι η Κομισιόν πρέπει να αποφασίσει αν θα παρέμβει ή όχι σε τέτοιες διαπραγματεύσεις. Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι όταν εμ, εμπίπτει, όταν πρόκειται για ευρωπαϊκές χώρες, θα πρέπει να συμμετέχει αυτόματα η Κομισιόν. Πρέπει να έχουμε κάποια οταν όμως. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να δεχτούμε ότι η Κομισιόν μπορεί να συμμετέχει με δική της πρωτοβουλία σε διαπραγματεύσεις ή όχι, αλλά όταν τη ζητήσει ένα κράτο μέλο θα πρέπει να είναι παρούσα στη διαπραγματεύση. Ένα τρίτο στοιχείο είναι ο πρώτερο έλεγχο τη συμβατότητα με προηγούμενε συμφωνίε. Που έχουν ήδη υπογραφεί δηλαδή. Κατά την άποψή μου αυτό ο εκ των προτέρων έλεγχο δεν θα πρέπει να γίνεται μόνο όταν το ζητά ένα κράτο μέλο, το οποίο έχει φτάσει πληροφόρηση, αν ο στόχος αυτής της ρήτρα είναι να μην συνάπτονται συμφωνίες οι οποίες θίγουν άλλα κράτη-μέλη, είναι λογικό ο έλεγχος αυτός να γίνεται και στην περίπτωση που η Κομισιόν έχει αποχρόντες λόγους για να θεωρήσει ότι η συμφωνία αυτή μπορεί να θίξει κάποιο άλλο κρατός μέλος. Ακόμα και αν τα εμπλεκόμενα κράτη-μέλη δεν έχουν ζητήσει να υπάρξει μια τέτοια αξιολόγηση συμβατότητος. Και τέλος, θα ήθελα να υπογραμμίσω και πάλι την ανάγκη <clears throat> να διευκρινίσουμε πλήρως τις ε, αρνητικής νομοδότησης για μια τέτοια συμφωνία από την ε, Κομισιόν. Αυτό ισοδυναμεί με μια αιτιολογημένη γνώμη που απευθύνεται σε μια χώρα για να καταλάβει η χώρα αυτή ότι εκθέτει τον εαυτό της ένα κίνδυνο και αν υπογράψει μια τέτοια συμφωνία μπορεί να, αυτό να οδηγήσει στην εκκίνηση μιας διαδικασίας επί παραβάση, εφόσον δεν θα δεχτεί την άποψη της Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Βιδάλ Κουάδρας. Έχουμε κλείσει τις παρεμβάσεις των ε, σκιωδών συγητών. Δίνω το λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν, εάν θέλει να λάβει το λόγο βέβαια. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με το ότι η Επιτροπή φαίνεται να στηρίζει την πρόταση της ε, Κομισιόν και την ενισχύει νομίζω κιόλας, είναι πολύ θετικό αυτό. Θα ήθελα να σχολιάσω κάποια πράγματα που αναφέρθηκαν ως σημεία κλειδιά, ξεκινώντα με τι εμπορικέ ε, συμβάσει. Εάν ένα κράτος μέλος στο πλαίσιο μια ε, διακυβερνητική συμφωνίας εκχωρήσει σε εμπορική εταιρεία το ρυθμιστικό πλαίσιο, ε, παραδείγματο χάρη στην περίπτωση ενός αγωγού, τα κράτη-μέλη μπορούν να ζητήσουν από την εταιρεία αυτή να μοιραστεί την εμπορική αυτή σύμβαση με τις αρχές. Και ακριβώς οι εμπορικές συμβάσεις που είναι μέρος διακυβερνητικής συμφωνίας είναι αυτές που πρέπει να δει η Κομισιόν για να κρίνει την συμβατότητα της συμφωνίας με το κοινοτικό δίκαιο. Αλλά βεβαίως ε, ε, οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικέ και προβλέπεται στην πρόταση της Κομισιόν πως τα κράτη-μέλη έχουν δικαίωμα να ενημερώσουν την Κομισιόν για τον βαθμό εμπιστευτικότητας ε, των πληροφοριών αυτών. Όσον αφορά τώρα το χρονοδιάγραμμα, να κάνω μια παρατήρηση για τη ρόλο παρατηρητού και την εξάντα αξιολόγηση των διακυβερνητικών συμφωνιών. Στόχος της συμφωνίας είναι να διασφαλίσουμε πως από νωρίς οι διακυβερνητικέ αυτέ συμφωνίε θα είναι συμβατέ με την νομοθεσία, την κοινοτική περιοριστική αγορά και την πολιτική ασφάλεια ενεργειακή. Αυτά μπορούν να διευκολυνθούν εάν η Κομισιόν είναι ενημερωμένη από την αρχή των διαπραγματεύσεων. Μοιραία, Βεβαίω, θα υπάρξει έτσι και η ανάγκη μιας αξιολόγησης εξάντε και θα μειώσουν και τον χρόνο αυτή τη αξιολόγηση. Εάν έχει λίγο χρόνο στη διάθεσή της η Κομισιόν για μια αξιολόγηση εξάντε, προφανώς η Κομισιόν δεν θα μπορέσει να δώσει μια οριστική απάντηση, αλλά θα πρέπει να θέσει όρους στην απάντησή της και αυτό δεν είναι προς το συμφέρον των κρατών μελών, επενδυτών ή καταναλωτών. Ένα τελευταίο σχόλιο για τις επενδυτικές συμφωνίες. Εάν υπάρχει ανάγκη να συμπεριληφθεί μία αναφορά προς το ότι θα εξεταστούν οι διμερείς επενδυτικές συμφωνίες για την συμμόρφωσή τους με την νομοθεσία εσωτερικής αγοράς, η αναφορά αυτή θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην, ε, στον κανονισμό της ε, διμερούς αυτής συμφωνίας και θεωρούν πως αυτό ισχύει ε, ιδιαίτερα ε, καθώς δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί αυτός ο κανονισμός και δεν μπορούμε να προδικάσουμε το αποτέλεσμα της διαδικασίας είναι απόφαση. Όπως ξέρετε, η πρόταση απόφαση περί διακυβερνητικών συμφωνιών περιλαμβάνει ήδη μια υποχρέωση αναφοράς προς την Κομισιόν και οι ε, διμερείς ενεργειακές συμφωνίες ε, που σχετίζονται με την ε, διακυβερνητική αυτή συμφωνία θα ληφθούν υπόψη. Αυτά και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο τελικός λόγος για τον κύριο Κάριντς. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Και αγαπητοί συνάδελφοι για τις ε, παρεμβάσεις σας. Ο λίγα σχόλια. Ως προς το πεδίο εφαρμογής Ασφαλώς θα πρέπει να το συζητήσουμε μεταξύ των σκιωδών, εάν δηλαδή θέλει το Κοινοβούλιο να προτείνει μια διακυβερνητική συμφωνία, μάλλον διακυβερνητική συμφωνία να καλύπτει και συμφωνία μεταξύ κράτους και ιδιωτικής εταιρείας. με ενδιαφέρει και αντιλαμβάνομαι αυτό που εννοούν οι συνάδελφοι. Μπορούμε να δούμε αν μπορούμε να καταφέρουμε να κερδίσουμε και το υπόλοιπο κοινοβούλιο. Εάν το κοινοβούλιο ακολουθήσει αυτή τη διατύπωση, σε μια καλή πλειοψηφία, σε μια ισχυρή πλειοψηφία, μπορώ να φανταστώ τι είδου αντιδράσει θα επιφυλάξουν ορισμένε χώρε, οι οποίε του ή είναι επιφυλακτικοί αντί αυτή συμφωνία. αλλά πάντω, ίσω και να μην είναι τόσο κακό αυτό, γιατί καλό είναι πότε πότε να είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα και οι θέσει. Θα το κοιτάξουμε. Βλέπω ποια ιδέα σας οδηγεί στις παρατηρήσεις αυτές. Αλλά ανεβάζει πολύ τις προσδοκίες ως προς το πεδίο εφαρμογής, ανεβάζει πολύ τον πύχη. Ε, ως προς την Ανάγκη για σαφήνεια που ανέφερε ο κ. Βιδάλ και βέβαια πρέπει να είναι σαφής η τροπολογία και προς το ενδεχόμενο μιας αρνητικής αξιολόγησης. Και πρέπει να προβλέπετε, και αυτό άλλωστε το έχω σε μια συμβαστική λύση, σκοπεύω να το περιλάω τουλάχιστον, σε μια συμβαστική τροπολογία, θα πρέπει σε περίπτωση που δεν λάβει υπόψη ε, την γνωμοδότηση αυτό το ε, κράτος μέλος και προχωρήσει η υπογραφή, τότε θα πρέπει να βλέπετε η εκκίνηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Διαδικασία σε παραβιάση ε, με την έννοια ότι μπορεί να μην είναι δεσμευτική η πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά εάν η Επιτροπή φρονεί ότι είναι αντίθετη με το κοινοτικό δίκαιο η παραγνώριση αυτή της πρόταση ίσω θα μπορούσε να προχωρήσει σε διαδικασία ε, παραβιάση. Από τους πράσινους και ίσως και από τους σοσιαλδημοκράτες ε, τέθη το ζήτημα των στόχων των ε, πολιτικών ενεργείας και για την κλιματική αλλαγή. Έχω και εγώ μια διατύπωση κάπως πιο ευρεία, Α το συζητήσουμε αύριο. Δεν έχω αντίρρηση προ τη βασική ιδέα. Ίσως το θεσίτημα είναι περισσότερο η ορολογία, η διατύπωση που θα ε, χρησιμοποιήσουμε και πώ θα αντικατοπτρίσει τη θέση του Κοινοβουλίου. Επίση, ε, ακούσαμε πει η Επιτροπή για τι συμφωνίε ω προ την επένδυση, τι επενδύσει. Α το ξανασυστήσουμε αύριο να δούμε αν μπορούμε να καταλήξουμε σε ε, συνένεση. Πέραν αυτού. Δεν νομίζω να ανέφερε κανείς άλλος τίποτα που να λησμόνησα. Πάντως και πάλι ευχαριστώ θερμά για την συζήτηση, για τις προτάσεις σας και αύριο με τους, με τους κοιόδες ηγητές θα τα πούμε πιο αναλυτικά. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Κάρνς, λέει η Πρόεδρος. Η ενδεικτική ψηφοφορία στην Ήτρε που θα δώσει και την εντολή για τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο 28 Φεβρουαρίου 2012. Και τώρα, τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Ανταγωνιστική ψηφιακή ενία αγορά, ήλε διακυβέρνηση ως καθοριστικός παράγοντας. Κυρία Τσίκα, όχι το λόγο. 45 λεπτά έχουμε στη μας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Μιλάμε για ηλεκτρονική διακυβέρνηση και μια ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά. Πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Η ψηφιακή ατζέντα είναι ουσιαστικό κομμάτι της στρατηγικής Ευρώπη. Οι 20, 20 υπάρχουν πολλές απόψεις. Θα προσπαθήσω όμως εγώ να κάνω μια σύντομη παρουσίαση του θέματος για να μπορέσουν και οι συνάδελφοι να λάβουν το λόγο γιατί θέλω να ακούσω τι άποψη έχουν. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω πως ένα σημαντικό στοιχείο της ημερήσιας διάταξης είναι οι τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για να υπάρχει, δυνατό, για να υπάρχει στον μεγαλύτερη καινοτομία. Η ψηφιακή ατζέντα προσφέρει διάφορες δυνατότητες στον τομέα των ε, ψηφιακών ε, κρατικών υπηρεσιών, π.χ. διασυνοριακές ηλεκτρονικές υπηρεσίες, η διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών κρατικών υπηρεσιών. έχει τη σημασία που έχουν ε, οι υπηρεσίες ε, μόνο απευθυντικές λεγόμενες, αλλά και οι ρύθμιση των ε, τεχνολογιών αυτών και η τυποποίησή τους τώρα. Από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν 20 διαφορετικά συστήματα, 12 απευθύνονται στους πολίτες, ε, πύχη, φόρος εισοδήματος, κοινωνικό σύστημα στήριξης, ε, άδειες οικοδομών, ε, ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες ε, και αλλαγή της ε, διεύθυνση διαμονής. Υπάρχουν κάποιες άλλες που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως ΦΠΑ, φόρος κύκλου εργασιών και τα λοιπά. Για να μπορέσουμε λοιπόν να Πρέπει να το χώρο αυτό των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Χρειάζεται ένα πλαίσιο και τέσσερα βήματα. Η δημοσίευση στο διαδίκτυο, το κατέβασμα ε, εντύπων ή και αμοιβαία λεπίδραση να συμπληρώνονται δηλαδή έγγραφα και το τελευταίο είναι συναλλαγές στο διαδίκτυο μεταξύ των οποίων και οι πληρώμες. Με βάση λοιπόν της νέας έκθεσης για τις ηλεκτρονικές τάσεις έχουμε αυτή τη στιγμή ένα 82% σε Αυστρία, Ιρλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία και Σουηδία όσον αφορά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και ε, φαίνεται πως αυτή τη στιγμή οι υπηρεσίες για επιχειρήσεις είναι πολύ πιο προχωρημένες από ότι οι υπηρεσίες για τους πολίτες και θα πρέπει να υπάρχει μία μοναδική υπηρεσία στην οποία να απευθύνει το πολίτη, όπω παραδείγματο χάρη στην Αυστρία, Δανία και Ηνωμένο Βασίλειο και θα δημιουργήσει νομίζω προσθέμενη αξία και αλλού. Τώρα για την πολυπλοκότητα των υπηρεσιών αυτών. Η Μάλτα, η Σλοβενία και δύο άλλες χώρε επίση νομίζω βρίσκονται στην πρώτη θέση. Το 2010 οι τοπικές αρχές είχαν μόνο ένα 50% των υπηρεσιών τους ε, στο διαδίκτυο. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καλύτερη διαλειτουργικότητα στον ευρωπαϊκό τομέα. Είναι το η ψηφιακή διαχείριση της ε, ταυτότητας ε, για να μπορέσει να λειτουργήσει πραγματικά η ψηφιακή υπηρεσία προς τον πολίτη και αυτό σημαίνει ως το επίπεδο της λειτουργικότητας πως όλες οι ηλεκτρονικές υπογραφές θα έπρεπε να μπορούν να αναγνωρίζονται και από άλλα κράτη-μέλη και άλλων, από άλλες υπηρεσίες πιστοποίησης δηλαδή. Αλλά βεβαίως ε, μέχρι στιγμής υπάρχει εμπιστοσύνη μόνο σε αυτά τα οποία πιστοποιούνται εντός του ιδίου ε, κράτους. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα πιστοποίησης ε, και φορέων υπηρεσιών που δεν είναι μόνο από την ίδια χώρα. Τα περισσότερα λοιπόν κράτη-μέλη έχουν ένα σύστημα ηλεκτρονικής υπογραφής ε, καθαρά εθνικό χωρίς να λαμβάνεται υπόψη πως ε, θα μπορούσαν να προσφέρονται τέτοιες υπηρεσίε και σε άλλα κράτη-μέλη. Δεν υπάρχει λοιπόν ένα πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως σας είπα, οι υπηρεσίε αυτές είναι προσανατολισμένες στο εθνικό. Θα ήθελα λοιπόν να προτείνω κάποια μέτρα στην έκθεσή μου, παραδείγματος χάρη Υπογραμμίζω πως δυστυχώς το 2011 μόνο ένα 50% των χρηστών χρησιμοποίησε έντυπα online. Δυστυχώς το διαδίκτυο δεν χρησιμοποιείται αρκετά, χρησιμοποιείται το κινητό διαδίκτυο, αλλά και οι επιχειρήσεις δεν χρησιμοποιούν αρκετά τις ε, υπηρεσίες αυτές. Θα πρέπει να υπάρχουν λοιπόν συστήματα ε, με καλύτερη πρόσβαση. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι πάρα πολύ σημαντική για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί έτσι μειώνεται το διοικητικό κόστος. Συχνά οι πολίτες και οι επιχειρήσεις ε, ε, αντιμετωπίζουν πάρα πολλά εμπόδια όταν προσπαθούν να δραστηριοποιηθούν σε αυτόν τον τομέα. Μεγάλα εμπόδια στο διασυνοριακό τομέα είναι η ηλεκτρονική πιστοποίηση και υπογραφή και η διαλειτουργικότητα η οποία ακόμα δεν υφίσταται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για να μπορέσουμε λοιπόν να έχουμε διασυνοριακές αποτελεσματικές υπηρεσίες στην Ένωση με διαλειτουργικότητα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις χρειάζεται ένα κοινό νομικό πλαίσιο το οποίο θα είναι σαφές και μια, ένα πλαίσιο αμοιβαίας αναγνώρισης των ηλεκτρονικών υπογραφών. Και βεβαίως το πρόγραμμα το πιλωτικό το οποίο υπάρχει για την διαλειτουργικότητα των διασυνοριακών υπηρεσιών. Καλούμε λοιπόν την Κομισιόν να επανεξετάσει το πλαίσιο και να μας πει εάν θα απαιτείται μία νέα οδηγία. Οι προδιαγραφές είναι πάρα πολύ σημαντικές και χαιρετίζουμε την ε, εντολή της Κομισιόν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Τυποποίησης για να οδηγηθούμε σε μία ευρωπαϊκή προδιαγραφή για την ηλεκτρονική υπόγραφη. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα διαλειτουργικότητας της λεγόμενης υποδομής private key και βεβαίως θα πρέπει να υπάρξουν και ευρωπαϊκά διοικητικά μέτρα σύμφωνα με το σχέδιο για το άνοιγμα της εσωτερικής αγοράς. Επίσης ζητάμε από τα κράτη-μέλη να καταστήσουν τις ε, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών πιο διάφανες και να δημιουργηθεί ένα σύστημα το οποίο θα ε, έχει στόχο την προστασία των κρίσιμων υποδομών στην Ευρώπη. Για τις δημόσιες προμήθειες να πω πως στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι δημόσιες δαπάνε αποτελούν 16% του ΑΕΠ, γι' αυτό ζητάμε οι ηλεκτρονικές δημόσιες προμήθειες να χρησιμοποιούνται μέχρι το 2015 για όλες τις ε, δημόσιες προμήθειες των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Επίσης ζητάμε το ίδιο να γίνει και για τις διάφορες άδειες και οι μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις να μπορούν να συμμετάσχουν στις ηλεκτρονικές αυτές δημοσιοπρομήθειες. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν δύο φάσεις, μία πρώτη και μία μετά την ε, απονομή της σύμβασης σε ε, κάποιον ανάδοχο, οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το έτος 2015. Όσον αφορά τώρα την τιμολόγηση, πρέπει να τονίσουμε πως η μέθοδος αυτή θα πρέπει να είναι σημαντικότερη μέχρι το 2020. Τονίζουμε επίσης πως η ηλεκτρονική τιμολόγηση έχει πάρα πολλά πλέον για τις πληρωμές, αυξάνεται η συλλογή του ΦΠΑ και είναι λιγότερο το διοικητικό κόστος. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει ίση αντιμετώπιση ε, από λογιστική σκοπιάς ε, χάρτινων και ηλεκτρονικών ε, τιμολογίων. Τονίζω επίσης πως Δανία, Φιλανδία, Ιταλία, Ισπανία και Σουηδία ήδη έχουν ένα τέτοιο εθνικό σύστημα λογιστικό όσον αφορά τις αρχές τους και ζητάμε να γίνει αυτό από όλες τις χώρες μέχρι το 2016. Τέλος θα πω πως όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ασχοληθούν με αυτό το θέμα και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως υπάρχουν και χρήστες οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ και θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να ε, γίνεται και με ε, χάρτινα έντυπα η όλη διαδικασία επίσης. Τα μέτρα της Κομισιόν περί ανοιχτών ε, δεδομένων εξακολουθούν να ισχύουν και θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν από τον δημόσιο τομέα. Τέλος, θα ήθελα να πω πως το Connecting Europe είναι ένα σημαντικό μέσο, 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ θα, θα επενδυθούν για την ευρυζωνικότητα. για πανευρωπαϊκά δίκτυα. Πρέπει λοιπόν να επεκτείνουμε αυτά τα δίκτυα και είναι σημαντικό τα κράτη-μέλη να προωθήσουν τις δομές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, να τις επεκτείνουν μάλλον σύμφωνα με το εθνικό και τα ευρωπαϊκά σχέδια δράσης. Η διαλειτουργικότητα λοιπόν πρέπει να αποτελέσει το σημείο εκείνο στο οποίο θα πρέπει να δώσουμε έμφαση και βεβαίω η άρχιση των προπολογισμών γι' αυτό. Σα ευχαριστώ. καλά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια κυρία Τικάου για την έκθεση που παρουσίασε, η οποία προσφέρει χρήσιμες θέσεις για την εξέταση αυτού του σημαντικού θέματος. Πρέπει να παραδειγματιστούμε από πράγματα που δεν πήγαν καλά σε όλες τις προηγούμενες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Πρέπει να θέσουμε έξυπνους και ευέλικτους στόχους που θα βοηθούν τα κράτη-μέλη που τώρα ξεκινούν την προσπάθειά τους, αλλά δεν θα εμποδίζουν όσους βρίσκονται ήδη μπροστά. Και ταυτόχρονα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε ένα κοινό επίπεδο πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που θα διασφαλίσουν μια ελάχιστη διαλειτουργικότητα ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η συγγήτρια κυρία Τικάου συνεισφέρει μερικές καλές προτάσεις για την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και άλλων ψηφιακών υπηρεσιών χρήσιμων για την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ενιαία ψηφιακή αγορά. Πιστεύω ότι είναι ένα καλό κείμενο βάσης, για το οποίο όμως υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης. Πολλές από τις προτάσεις της κυρίας Τικάου βρίσκονται σε απόλυτη ταύτιση με τους τεθέντες στόχους της ψηφιακής ατζέντα. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να ταιριάξουμε ακόμα καλύτερα το κείμενο της Επιτροπής Ήτρε με την ευρωπαϊκή αυτή εμβληματική πρωτοβουλία. Επίσης, σε αρκετά σημεία η κυρία Τικάο υποκύπτει στον πειρασμό να προτείνει τεχνικές λύσεις για e-government, e-invoice, η identity και ούτω καθεξής. Πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε η Επιτροπή Ήτρε να υποδεικνύει λύσεις στους ειδικού. Δεν είναι δική μας δουλειά. Θα έπρεπε να έχουμε μια τεχνολογικά ουδέτερη προσέγγιση. Έχουμε σκοπό να καταθέσουμε μια σειρά από τροπολογίε σε συμφωνία με τις πάγιες πολιτικές γραμμές του ΕΛΚ. Θα θέλαμε, παραδείγματο χάρη, περισσότερη ευελιξία για τις κυβερνήσεις, για τους εθνικούς στόχους που θέτουν και τους τρόπους με τους οποίους τους υλοποιούν. Περισσότερα κίνητρα για τον ιδιωτικό τομέα και τη σύνδεση δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Μεγαλύτερη υποστήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και προβλέψεις για την ενίσχυση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας το e-government είναι ένας κλάδος με μεγάλη οικονομική σημασία τόσο για τον δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει να σημειώσω ότι ιδιαίτερα για τα κράτη-μέλη που πλήττονται από την κρίση όπως στη δική μου χώρα η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι μια ιδανική λύση για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, ενίσχυση της παραγωγικότητας και προώθηση της διαφάνειας. Ανεξάρτητα από την κατάσταση μιας χώρας, ως προς την πρόοδο της σχετικά με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, το e-government πρέπει να προωθηθεί και να εφαρμοστεί, καθώς οι προηγμένες υπηρεσίες τεχνολογιών παρέχουν νέες τεράστιες ευκαιρίες για τη βελτίωση των δημοσίων υπηρεσιών για τους πολίτες και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των κυβερνητικών ενεργειών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Πρόεδρο. Θέλω και εγώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς την <coughs> εισηγήτρια για την τόσο ενδιαφέρουσα αυτή η έκθεση. Θα ήθελα τώρα να προσθέσω και κάποιες νέες προτάσεις σε αυτή την πρόταση η Σλοβενία από την οποία έλκω την καταγωγή, πριν από ορισμένα χρόνια είχε την πρωτοπορία στην Ευρώπη και πήρε και βραβείο σχετικά για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Ο στόχος μας ήταν να υπάρξει μια ελευθερία ροής όλων αυτών των στοιχείων, αλλά αυτό είναι δυνατό μονάχα άμα υπάρξει η δημιουργία των προϋποθέσεων για την κυκλοφορία αυτών των πληροφοριών. Το πιο σημαντικό είναι <clears throat> να υπάρξει η δυνατότητα πληροφόρησης εκ των άνω προς τα κάτω. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν ε, αυτό να αναπτυχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εκ των κάτω προς τα άνω. Μπορούμε λοιπόν έτσι με την ε, δημιουργία υπηρεσιών χάρη στην ηλεκτρονική τεχνολογία να βελτιώσουμε πολύ την κατάσταση στην κυβέρνηση. Ευχαριστώ πολύ. Τέλεια, τέλεια λέει η πρόεδρο. Μάλιστα έχετε το λόγο. Ο κύριο Κέλλη. Θα είμαι σύντομος κυρία Πρόεδρε, θέλω να πω απλώς ότι υποστηρίζω κατά 100% αυτή την πρόταση για την ηλεκτρονική ανάπτυξη της Ευρώπης, όλα αυτά που έχουν να κάνουν με ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονική ανάπτυξη, ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική κυβέρνηση. Όλα αυτά τα υποστηρίζω. Εγώ είμαι πολύ μέσα στα ηλεκτρονικά και τονίζω ότι είναι επιτέλους καιρός να πείσουμε τους νέους και όλους τους αυτούς που μπαίνουν στον τομέα το διακυβερνητικό να παράγουν υπηρεσίες οι οποίες θα είναι επιγραμμικά προσβάσιμες ώστε σε 4-5 ε, χρόνια να μπορούμε να έχουμε μια επαναστατικού χαρακτήρα ανάπτυξη στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και υπηρεσίες. Και λάβουμε υπόψη και την οικονομική κατάσταση και το δυναμικό στο ηλεκτρονικό εμπόριο το οποίο διαγράφεται προς το παρόν μόνο 75% των ηλεκτρονικών αυτών εταιριών ε, περιορίζονται στο δικό τους κράτος μέρος και τα 85% αυτών των εταιριών δεν ξεπερνούν τα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε είναι απαραίτητο να δημιουργήσουμε μια μεγαλύτερη ανάπτυξη αυτών των υπηρεσιών και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προωθήσουμε αυτή την πορεία και αυτή την τάση. Ευχαριστώ, λέει η Η Κομισιόν. Ευχαριστούμε. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το σχέδιο έκθεση. Νομίζω πως κατάφερε να μεταφέρει σε 13 σελίδες αριστουργηματικά ένα θέμα το οποίο είναι τόσο ευρύ όσο η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Εγώ θα περιοριστώ στο κομμάτι του σχεδίου δράσης περί ηλεκτρονικής ε, διοίκησης. Καλωσορίζουμε την γνωμοδότηση αυτή αξίζει, με συγχωρείτε, αγγίζει τις ε, βασικές πτυχές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αλλά και της ολοκλήρωσης της εσωτερικής ψηφιακής αγοράς και άρα ευπρόσδεκτη άποψη της ηγήτριας για την ε, ανάγκη που υπάρχει για μια ολοκληρωμένη άποψη για την ηλεκτρονική υπογραφή, την ηλεκτρονική ταυτότητα. Η Κομισιόν αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται πρόταση κανονισμού που μέχρι το τέλος της άνοιξης θα είναι έτοιμη. Θεωρούμε επίσης πως ε, πρόκειται για τον τομέα κλειδί για να μπορέσουν όλοι να υποφεληθούν από την ηλεκτρονική διοίκηση. Δικαίως λέτε πως είναι καλή για τις επιχειρήσεις, για τους πολίτες και για τη δημόσια διοίκηση. Αλλά χωρίς ε, ηλεκτρονική ταυτότητα, ταυτοποίηση, αυτό δεν γίνεται. Και η ανάγκη ε, αμοιβαία αναγνώριση αυτών των συστημάτων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωση. Ε, δυνατή την ενιαία αγορά. Επίσης για τις ηλεκτρονικές δημόσιες προμήθειες βεβαίως είναι κάτι το απολύτω απαραίτητο αυτό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα έχουμε έτσι διαφάνεια, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, χαμηλότερο κόστος και είναι κρίσιμο για την ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Θα ήθελα τέλος να πω πως η προσέγγιση που βλέπουμε στο σχέδιο αυτό της έκθεσης ε, λίγο πολύ κινείται στις κατευθύνσεις του σχεδίου δράσης του δικού μας και της ψηφιακής ατζέντα για την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Και τώρα ρωτάω αν, ζητά, θέλει να πει κάτι ακόμη η συγγήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που έλεγαν το λόγο και, και να επισημάνω ότι όπως είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχουν ακόμη κάποια εμπόδια ως προς τις εκθέσεις μας έχουμε περιορισμό και δεν μπορούμε να επεξεργαστούμε τα θέματα όπως θα θέλαμε και όπως θα έπρεπε. Θα ήθελα λοιπόν να υπογραμμίσω ότι οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες, η ηλεκτρονική ατζέντα έχουν μεγάλη σημασία και πρέπει να αποκτήσουν μεγάλη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επί παραδείγματι, επιχείρηση από τη Γαλλία σήμερα δεν θα ήταν σε θέση να συμμετάσχει σε ένα διαγωνισμό στη Βουλγαρία. γιατί δεν υπάρχει διαλειτουργικότητα, αμοιβαία αναγνώριση δηλαδή τη ηλεκτρονική υπογραφή, Λόγω αυτή τη απουσίας αναγνώριση, δεν θα μπορούσε να συμμετάσχει. Και άλλε τεχνικοί φραγμοί ήδη εμπόδια υπάρχουν βεβαίω, αλλά υπάρχουν πάνω από όλα αυτή οι διοικητική φραγμή, αυτέ οι διοικητικέ δυσκολίε που θα πρέπει να εξαλειφθούν. Μια πρώτη προσπάθεια γίνεται με αυτή την οδηγία λοιπόν με την μονοθυριδική προσέγγιση για το 2010 όπως προβλεπόταν στην προσφορά ε, ηλεκτρονικών υπηρεσιών ε, στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους. Ωστόσο δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όπως υπόθηκε και νωρίτερα. Έχουμε να κάνουμε μια προσέγγιση που δεν μπορεί να επιβληθεί άνωθεν μόνο. Πρέπει να ξεκινήσει και από τη βάση η προσπάθεια και ο κάθε εμπλεκόμενος να σε θέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικά. Βεβαίως θα πρέπει να προσφέρονται και σε ηλεκτρονικό επίπεδο οι σχετικές υπηρεσίες από τις τοπικές αρχές και να υπάρχει δυνατότητα εάν κάποιος θέλει Φερρυπίν ε, να ε, πάει σε ένα άλλο κράτος για να συνεχίσει τις σπουδές του. Ε, να είναι σε θέση να διατηρήσει την επαφή του με τα ηλεκτρονικά μέσα, με τις αρχές της πατρίδας του, Φερρυπίν, ε, εφορίες και ούτω καθεξής. Αυτό είναι μια βασική υπηρεσία που μπορούμε να προσφέρουμε στον πολίτη. Μπορούμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε αυτή την ψηφιακή ενιαία αγορά. Ο ρόλος των αρχών είναι πολύ σημαντικός, πρέπει να δώσουν το καλό παράδειγμα πάνω απ' όλα και στο ηλεκτρονικό εμπόριο ένα πολύ καλό παράδειγμα που θα ήθελα να επισημάνω είναι το, η δυνατότητα για υποβολή, για ανακήρυξη, προκήρυξη και συμμετοχή σε ε, διαγωνισμούς δημοσίων προμηθειών με τα ηλεκτρονικά μέσα που εξασφαλίζουν, ε, ταυτόχρονα σαν δυνατότητα και μεγάλη διαφάνεια. Ε, χώρες οι οποίες εισήγαγαν το σύστημα αυτό σε διάφορες κατηγορίες εμπορευμάτων, προϊόντων, ε, κατάφεραν σημαντική μείωση της δαπάνης τους, χάρη ακριβώς στην ηλεκτρονική προκήρυξη, τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Αυτό πιστεύω απαιτείται να προωθηθεί ταχύτατα. Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα να μπορούν να προσφέρονται από οποιοδήποτε κράτος σε οποιοδήποτε κράτος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έτσι πιστεύω ότι και βεβαίως η ε, τα ποσά που έχει προπολογίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν πολύ μεγάλη σημασία, το Connecting Europe, αλλά και πολλές άλλες δραστηριότητες μπορούν να βοηθήσουν, όπως το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα στο 2020 ή οι εθνικοί προϋπολογισμοί που μπορούν να στηρίξουν τέτοιες ε, πρωτοβουλίες. Επίσης η, πρωτοβουλία, η ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών του δημοσίου τομέα, των δημοσίων δηλαδή υπηρεσιών, που μπορούν να διευκολύνουν καταρχάς τον ε, πολίτη στο ιστορικό της χώρας, αλλά και δευτερευόντως ε, εκτός αυτής. Ευχαριστώ πολύ όλους τους αδέλφους όσοι έλαβαν το λόγο και θεωρώ όντω ότι χρειάζεται μια βελτίωση το κείμενο αυτό. Περιμένω να δω τις τροπολογίες σας, γιατί είμαι πεπισμένη ότι μπορούμε με την έκθεση αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ε, σηματοδοτήσουμε ε, τις εξελίξεις στον τομέα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Ε, σας ευχαριστώ για τα συμπεράσματά σας αυτά τροπολογίες μέχρι την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 12 η ώρα. Είναι η προθεσμία. Οι επόμενες συνεδριάσεις επιτροπής μας προβλέπονται για τις 27 Φεβρουαρίου 3 με 6.30 και 28 Φεβρουαρίου από τις 9 μέχρι τις 6.30. Εξαντλήσαμε τα σημεία της ημερήσιας διάταξης. Λίγη λοιπόν η συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.